Ε, Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήλθατε στη συνεδρίασή μα και καλημέρα. Για τη συνεδρίασή μα θα λάβει χώρα σήμερα σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα. Φαντάζομαι δεν έχετε παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη ούτε για τα πρακτικά των προηγουμένων μας συνεδριάσεων. Όλα αυτά στη διάθεσή σας. Εάν δεν έχετε καμία αντίρρηση θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί. Θα ξεκινήσουμε με μια ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Πολιτικών Αεροσκαφών. Είναι ένα θέμα που είναι επίκαιρο από πολλές απόψεις. Έχει μόλις ε, λάβει χώρα το, σαλόνι του, το αεροναυτικό σαλόνι του Μπουρζέ στο Παρίσι που είναι μια μεγάλη εκδήλωση μια μεγάλη έκθεση σε παγκόσμιο επίπεδο που αφορά τον αεροδιαστημικό χώρο και φέτος παρά τις δυσμενείς ε, μετεωρολογικές ε, ε, συνθήκες και παρά την, ε, τις δυσκολίες που είχε σε επίπεδο επικοινωνιών, τηλεφωνίας κυρίως, είχε μεγάλη επιτυχία. Αλλά πέραν του σαλονιού του Μπουζέ, μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό λόγω και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, μάλλον του που θα ασχοληθεί με θέματα άμυνας και ασφάλεια στο τέλος του έτους και μέσα στα οποία περιλαμβάνονται τα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας. Η αμυντική βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό επικαλύπτεται με την αεροναυτική βιομηχανία. Είναι ένα από τα κλειδιά αυτή η βιομηχανία της ε, ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης σε ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα και φυσικά η απώλεια αυτού του σημαντικού κρίκου της αεροναυτικής βιομηχανίας έχει σοβαρές συνέπειες. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές οι ανησυχίες που διατυπώνονται σε ευρύ επίπεδο για την σταδιακή απώλεια τεχνολογικής ικανότητας, ακόμα και ενδεχομένω πολιτικής θέλησης των Ευρωπαίων, για να έχουν μια υψηλού επίπεδου πολεμική αεροπορία στο μέλλον. Προφανώς όλα αυτά είναι πολύ γιατί από τεχνολογική άποψη είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου όλα αυτά τα ζητήματα αλλά έχουμε διαπιστώσει την χρησιμότητα αυτής της ε, αεροπορίας τις δύο τελευταίες συγκρούσεις οποίες ενεπλάκησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Λιβύη και στο Μαλί όπου η αεροπορία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σίγουρα στην περίπτωση της Λιβύης, αλλά επίσης και σε ό,τι αφορά στις ε, επιχειρήσεις στο Μαλί. Αυτή λοιπόν η ικανότητα της ε, αεροπορίας, της πολεμικής αεροπορίας, δυστυχώς δεν είναι κάτι το αυτονόητο, διότι απαιτούνται επενδύσεις, απαιτείται πολιτική θέληση, εκτός εάν θέλουμε η Ευρώπη να χάσει την ικανότητά της στα θέματα αυτά. Για να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε <clears throat> εξέχοντα μέλη του αεροναυτικού χώρου που θα μας παρουσιάσουν το έργο της Ακαδημίας Αεροσκεδιαστήματος της Τουλούζης. Αυτή είναι μια γαλλική ακαδημία αλλά η οποία έχει ιδιαίτερα ευρωπαϊκό χαρακτήρα και βασίζεται στην Τουλούζη. Είναι τρισιδική ο στρατηγός Μπρεβό ο οποίος έχει μια μακρά καριέρα στην αεροπορία, πολεμική αεροπορία και ο οποίος έχει εργαστεί και στην αερο... αεροναυτική βιομηχανία, τον κύριο David Marshall, ο οποίος επίσης έχει μία μακρά καριέρα στη Rolls Royce και είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αεροστη... Αεροδιαστημικών Εταιριών και τον κύριο Μπριντέλ, ο οποίος και αυτός ε, έχει περάσει μεγάλο διάστημα σε αυτή την Ακαδημία και είναι επικεφαλής μιας εταιρείας αεροναυτικής. Θα δώσω λοιπόν καταρχήν το λόγο στον στρατηγό Μπρεβό και μετά στους επόμενους ομιλητές. Στρατηγέ μου έχετε το λόγο. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καλαθάς εξ ονόματος των συναδέλφων μου να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να προβούμε σε αυτή την ανταλλαγή των απόψεων σε ό,τι αφορά την ε, πολεμική αεροπορία για ένα θέμα που κατά την άποψή μας είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Γιατί είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Γιατί η Ευρώπη, λόγω των αποφάσεων που ελήφθησαν στο παρελθόν, έχει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Πράγματι έχει μια πολεμική βιομηχανία η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και η οποία επανδρώνει ένα κλάδο που είναι ιδιαίτερα ικανός όπως αποδείχτηκε από τις πρόσφαρες συνταγηράξεις. Αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος να εξαφανιστεί στο μέλλον. Υπάρχει ο κίνδυνος και να πεθάνει, να εξαφανιστεί λόγω απουσίας αποφάσεων που θα έπρεπε να ληφθούν σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολεμικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα από ουσία αποφάσεων που αφορούν τη μελλοντική γενεά. Οι, απο... Οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές και από στρατηγική και από πολιτική άποψη. Μια τέτοια εξαφάνιση δεν θα έχει μόνο βιομηχανικές <clears throat> και πρακτικές επιπτώσεις μετά από 20 χρόνια ενδεχομένως θα, σταθούμε μάρτυρες μιας υποβάθμισης της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα. Για τον λόγο αυτό ακριβώς κρίναμε ότι ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα μπροστά σας, λαμβάνοντας υπόψη την βαρύτητά του. Η Ακαδημία είναι ένας οργανισμός ευρωπαϊκού χαρακτήρα και εξέφρασε και στο παρελθόν ε, την ανησυχία της για τον κίνδυνο αυτό που υπάρχει και συνεπώς κινητοποιήθηκε ως προς το θέμα αυτό. Εδώ και ένα χρόνο ασχολούται με, ασχολείται με μία μελέτη, το 2001 εξέδωσε ένα έγγραφο το οποίο μπορείτε να βρείτε στα έγγραφα που σας έχουν διανεμηθεί. Μετά η Ακαδημία οργάνωσε μία συνάντηση για το θέμα αυτό το Μάιο του 2013. Το φόρουμ αυτό επιβεβαίωσε τους φόβους μας, αλλά παράλληλα μας επέτρεψε να υποβάλουμε προτάσεις και να προτείνουμε λύσεις. Θα ήθελα να προτείνω για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα όσα σκοπεύουμε να πούμε ότι το θέμα αυτό αφορά αεροσκάφη χωρίς χειριστή και αεροσκάφη με χειριστή. Για τι θέμα πρόκειται. Με τη Όλες οι πρόσφατες σειράξεις, όλες και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, μας δείχνουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια βιομηχανία υψηλής απόδοσης. Αυτό είναι το νουκάνευ για να υπάρχει κυριαρχία, γιατί αυτό οδηγεί στη νίκη και στην λήψη των αποφάσεων. Τρία παραδείγματα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης στο κοσυφοπέδιο, το γεγονός και μόνο ότι ε, αναπτύχθηκε σαν δράση, επέτρεψε να ληφθούν αποφάσεις και μπόρεσαν να επιστρέψουν τα στρατεύματα χωρίς απώλειες. Στην Λιβύη, στο Μαλί, η ε, πολεμική αεροπορία έδειξε μία ικανότητα να διαδραματίζει βασικό ρόλο. Ενώ υπάρχουν ακόμα απειλές στις ε, περιοχές που πλήττονται από την κρίση, τα ευρωπαϊκά ε, αεροσκάφη μπόρεσαν να κινητοποιηθούν άμεσα. Αυτό δείχνει τις ε, αρετές αυτού του κλάδου. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα παρέμβασης εξουδετερώσης του αντιπάλου. Επιτρέψτε μου να παραθέσω ένα παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Μαλί, η πρώτη αποστολή που έγινε έδειξε τις δυνατότητές της γιατί ε, επανέβησε σε 9 και 45 και στην πρώτη κιόλας αποστολή κατέστρε, κατάφερε να καταστρέψει 21 στόχους. Καταφέρνει να έχει απόλυτο έλεγχο, να είναι ακριβής γιατί αυτό επιτρέπει την ε, αποφυγή των παράπλευρων απολειών και δυνατότητα επαναφοράς. Ε, βλέπετε ότι πλήττει άμεσα το στόχο της και με μεγάλη ακρίβεια. Αυτή η ικανότητα είναι κάτι που κατέχει η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει την ε, τρίχη να νίκει στις χώρες αυτές που έχουν τη δυνατότητα να συλλαμβάνουν, να αναπτύσσουν, να παράγουν μαχητικά αεροσκάφη, γιατί ε, έχει τεχνολογία υψηλού επίπεδου έχει ε, παράγει και είναι ε, μαχητικά τρία αεροσκάφη, Ιροφάν και Αεροφάν και Είναι ε, πραγματικά και τα τρία πάρα πολύ εντυπωσιακά και κατάφεραν να δείξουν τις δυνατότητές τους. Αυτή τους η ικανότητα είναι ανεξάρτητη, ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός Ευρώπη και αυτό αποτελεί στρατηγικό και πολιτικό πλεονέκτημα μεγάλης βαρύτητας. Δυστυχώς, αυτό το βασικό πλεονέκτημα που έχουμε την τύχη να διαθέτουμε γιατί ε, έχουν ληφθεί αποφάσεις σε έθετο χρόνο, υπάρχει περίπτωση να πάψουμε να το έχουμε γιατί δεν λαμβάνονται αποφάσεις την επόμενη γενιά. Κατά την άποψή μας ήταν κάτι καταστροφικό από άποψη στρατηγική και αν εγκαταλείψουμε αυτή την ικανότητα δεν θα καταφέρουμε ποτέ να τη βρούμε <clears throat> ξανά. Πώς έχουν τα πράγματα στις άλλες χώρες του κόσμου. Οι Αμερικανοί, όπως ενδεχομένω γνωρίζετε, έχουν ήδη ένα σκάφος τρίτης γενεάς, το F-22, και αναπτύσσουν, έχοντας πάρει ένα μέρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού, το F-35. Με δυσκολίες ε, βεβαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν να κάνουμε με ένα αεροσκάφος της νέας γενεάς. Ακόμα πιο σημαντικό και ακόμα πιο σοβαρό, οι αναδυόμενες χώρες, οι επαναναδυόμενες, κατάλαβαν καλά ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας λυσαλέας μάχης σε επίπεδο τεχνολογίας. Ε, αυτό συμβαίνει στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ινδία, στην ε, ε, Νότια Κορέα. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν ε, αντιδρά σε αυτό το τομέα. Τώρα, για να μπορέσουμε να επισέλθουμε περισσότερο σε επιμέρους θέματα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου από την Ακαδημία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζωσέ που θα μας μιλήσει για την παρούσα κατάσταση. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Α, Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου από το πρίσμα της βιομηχανίας και όπως τα καταλαβαίνετε και από την προφορά μου είμαι Ελβετός αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της σταδιοδρομίας μου ε, υπήρξε στο εξωτερικό. Ο στρατηγός Μπρεβού σας εξήγησε ήδη περί τίνος ακριβώς πρόκειται σε επίπεδο στρατηγικής. Πολύ σύντομα λοιπόν θα μου επιτρέψετε να επανέλθω και εγώ στη νέα γενιά των μαχητικών αεροσκαφών. Οποτεδήποτε αναφέρουμε τα μαχητικά αεροσκάφη, είτε είναι πανδρομένα είτε όχι, υπάρχει πάντα ο χειριστής, είτε βρίσκεται μέσα στο αεροσκάφος είτε όχι. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη, κυρίως ε, στην Κίνα, που αφορά σε δύο γνωστά αεροσκάφη, το 20 και 23, στη Ρωσία το T50, από κοινού κατασκευάστηκε αυτό με την ε, Κίνα, στην ε, Κορέα, στην ε, Τουρκία. Υπάρχουν νέα μοντέλα αεροσκαφών όπου ο εφοδιασμός γίνεται στον αέρα και κατόπιν τούτου μπορούν να έχουν άλλη εμβέλεια. Αυτά σύντομα θα εμφανιστούν στην αγορά και θα μπορούν και να εξάγονται. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς ε, ως Ευρωπαίοι οφείλουμε να τα λάβουμε υπόψη μας. Ε, όσον αφορά το φόρουμ ε, στο Παρίσι που αναφέρθηκε επίσης από τον προλαλήσαντα, στο φόρουμ αυτό γνωστοποιήθηκαν διάφορα προγράμματα από την Ευρώπη δεν είναι δηλαδή αλήθεια ότι δεν γίνεται τίποτα. Υπήρχαν κάποια προγράμματα επίδειξη. και αυτό όμω που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα διάσπαρτο. Δηλαδή λαμβάνουν χώρα παράλληλες ε, δραστηριότητε. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη γραμμή και πλέψη όσον αφορά το ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Έχουμε την τεχνολογία η οποία σε μεγάλο βαθμό προάγεται μέσα από συνεργασίες. Όσον αφορά την ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, στην ΕΝΤΑ υπάρχουν προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει και εγώ. Προγράμματα που οργάνωσε η Γερμανία που στέφτηκαν από ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά τα προγράμματα αυτά ε, που αφορούν το 10-15% δεν επαρκούν, τουλάχιστον όσον αφορά την Ευρώπη. Κατά τα άλλα, στο φόρουμ αλλά και στη δική μας γνωμοδότηση του 2011 καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν μεν δύο τομείς ε, Υπάρχουν μάλλον δύο τομείς που δημιουργούν προβλήματα. Ο ένας τομέας είναι η δική μας η δυνατότητα να κατασκευάζουμε μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφοράς. Ε, εκεί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και έχουν ήδη αναφερθεί. Όσον αφορά τη συμβατική τεχνολογία, αυτή πρέπει να είναι επαρκής να έχουμε προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο και αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν δυνατότητες και τεχνολογίες οι οποίες λόγω των απαιτήσεων εμφανίζονται όλο και περισσότερο. Υπάρχουν αισθητήρε, υπάρχουν τα link σε δεδομένα, η διαδικτύωση, γιατί ξέρετε στον τομέα των, των μαχητικών αεροσκαφών δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τη διαδικτύωση ανάμεσα σε διάφορους εμπλεκόμενους. Δηλαδή η διαδικτύωση δεν γίνεται μόνο και δεν έχει σημασία σημασία μόνο ανάμεσα στα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά προφανώς και με τις βάσεις εδάφους. Αυτό λοιπόν απαιτεί ε, νέα τεχνολογία. Και γενικά όσον αφορά την εξέλιξη της ε, τεχνολογίας και την δυνατότητα διατήρησης της απόδοσης, προφανώς και εμφανίζεται πίεση για εξορθολογισμό. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα κονδύλια εκ των προτέρων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δείξουμε πώς τα κονδύλια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που θα συζητήσουμε και αργότερα. Θα ήθελα τώρα να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου, τον David Marshall, ο οποίος θα μιλήσει για την βιομηχανική βάση. Thank you, George, Uh, Ευχαριστώ πολύ, <coughs> το τμήμα το οποίο θέλω να καλύψω προσωπικά είναι το θέμα της σημασίας της ύπαρξης μιας βιομηχανικής βάσης στον αεροναυτικό τομέα για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε επιχειρήσεις και για να μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό στα θέματα αυτά. Μπορεί να μην γνωρίζετε το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι στρατιωτικές δυνάμεις σε όλες τις χώρες του κόσμου χρησιμοποιούν τη βιομηχανία για κάθε επίπεδο υποστήριξης του εξοπλισμού τους. Αυτό περιλαμβάνει και τις επιχείρησεις, τις στρατιωτικές επιχείρησεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι μία από τις ηγετικές χώρες στα θέματα αυτά. Και όλα τα μεταγωγικά αεροπλάνα και τα αεροπλάνα Tiger στο Νόρτον της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας υποστηρίζονται από τη βιομηχανία και πηγαίνουν εκεί όπως όταν είναι απαραίτητο για επισκευές και ελέγχους. Και στο, και στο Μόρον γίνεται το ίδιο πράγμα για τα Tornadoes, τα οποία επίσης είναι τα, όπως γνωρίζετε, είναι τα βασικά αεροπλάνα κρούσης του Ηνωμένου Βασιλείου στις στρατιωτικές τώρα επιχειρήσεις. Αυτό αρχίζει να γίνεται ένα πάρα πολύ επίκαιρο και συχνό θέμα. Υπάρχει μια ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι λεγόμενες κατεπίγουσες επιχειρησιακές ανάγκες. Δηλαδή σε μια κατάσταση εμπόλεμη, όταν ανακαλύψει η μαχητική δύναμη ότι χρειάζονται να γίνουν κάποιοι, κάποιες μεταλλαγές στον εξοπλισμό της, ε, μετά από την χρήση των αεροσκαφών, και χρειάζεται να γίνει πολύ γρήγορα αυτή η αναβάθμιση των μαχητικών ικανοτήτων των αεροσκαφών. Αυτό απαιτεί μια ε, βιομηχανία η οποία μπορεί να είναι έτοιμη και έχει την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να κάνει αυτές τις αναβαθμίσεις. Όταν λέω ότι έχει την τεχνογνωσία εννοώ να μπορεί να ξέρει τι χρειάζεται για να κάνει αυτή την αναβάθμιση, επομένως να ξέρει πώς έχει σχεδιαστεί το αεροπλάνο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Τώρα, σε μια άλλη χώρα, φυσικά αυτές οι πληροφορίες δεν είναι εύκολο να τις αποκτήσει κανείς. Μπορεί κανείς να τις έχει ή να μην τις έχει και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να κάνει κανείς αυτή την αναβάθμιση χωρίς να ξέρει αυτές τις πληροφορίες. Επομένως η ίδια η ικανότητα που έχει μια βιομηχανική μονάδα για να προχωρήσει σε αυτές τις αναβαθμίσεις παίζει σημαντικό ρόλο στη νίκη σε πολεμικές συγκρούσεις. Έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα στη Γερμανία όπου το Global Hawk, τα μη επαντρωμένα αεροπλάνα τα οποία είχαν αγοράσει, αναγκαστήκαν τελικά να ε, ακυρώσουν το συμβόλαιο γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τις ΗΠΑ τα απαραίτητα στοιχεία για να αναβαθμίσουν αυτά τα αεροσκάφη και το κόστος του να πάρουν αυτά τα στοιχεία ακόμα και αν μπορούσαν θα ήταν απαγορευτικό. Και αυτό ήταν πρόσφατο γεγονός, ήταν κάτι που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα είναι επίκαιρο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά την διατήρηση της ικανότητας και βιομηχανικής βάσης για τα αεροσκάφη αυτά. Μια άλλη πτυχή της ε, βιομηχανικής βάσης είναι ότι ο τομέας αυτός της βιομηχανίας αποτελεί και ένα κινητήριο μοχλό και υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια για την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και φυσικά απαιτεί και υψηλά προσοντούχους εργαζόμενους, όχι μόνο για το δικό του το τομέα, αλλά και για τους συναφείς τομείς και για την αεροδιαστημικό τομέα και άλλους τομείς. Πρέπει να σκεφτείτε ότι η χρονική κλίμακα για την ανάπτυξη νέων αεροσκαφών είναι της τάξης των 20 ετών από τον αρχικό σχεδιασμό με την επιχειρησιακή ικανότητα. Έχουμε τα αεροπλάνα όπως είναι το Ρήπον, το Ραφάλ, γιατί πήραμε πριν από 20 χρόνια τις απαραίτητες αποφάσεις που μας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε την τεχνολογική ικανότητα και να αναπτύξουμε αυτή την τεχνολογική ικανότητα για να φτάσουμε σε λειτουργικά αεροσκάφη. Οι επιχειρησιακές ανάγκες <clears throat> για ένα μαχητικό αεροσκάφος βρίσκονται <clears throat> στην αιχμή της λόγχης της ε, τεχνολογικής ικανότητας. Ζητούμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση και την μεγαλύτερη ικανότητα των αεροσκαφών για να κερδίσουμε μάχες. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η τεχνολογία αιχμής έρχεται πάντα από τον αεροναυτικό βιομηχανικό τομέα. Σκεφτείτε την ε, τουρμπίνα ε, μιας ενός κινητήρα αεροσκάφους, τις ε, πάλες της ε, τουρμπίνας που ουσιαστικά λειτουργούν πάνω από το σημείο τήξης του μετάλλου από το οποίο αποτελούνται αυτές οι λεπίδες και αυτό γίνεται χάρη σε μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη τεχνολογία ψήξης που χαμηλώνει την θερμοκρασία. Και αυτό χάρη σε μια στρατιωτική τεχνολογία που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Το fly-by-wire είναι μια επίση πολύ σημαντική τεχνολογία που ξεκίνησε στο στρατιωτικό τομέα και τώρα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και στα εμπορικά αεροσκάφη. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να σα πω ότι έχουμε τα έρμπα στα οποία είναι τόσο επιτυχή γιατί προηγουμένως υπήρξε η στρατιωτική τεχνολογία η οποία μεταλαμπαδεύτηκε στα εμπορικά αεροσκάφη. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχίσει στο μέλλον και ακόμα και τώρα μπορούμε να διαβλέψουμε τη μορφή που θα έχουν τα μελλοντικά αεροσκάφη στον εμπορικό χώρο που θα εξαρτώνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο στρατιωτικό τομέα που τώρα εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι απαραίτητες. Τα λεγόμενα απόλυτα ηλεκτρικά αεροσκάφη που, όπου δημιουργείται πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στο αεροσκάφος και διανέμεται σε όλο το αεροσκάφος, αυτό μπορεί να είναι κομβικού χαρακτήρα για τα μελλοντικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μαχητικού χαρακτήρα και αυτό αναφέρεται ήδη από την Airbus ως μια πιθανή επιλογή για τη μελλοντική γενιά εμπορικών αεροσκαφών. Εάν δεν προχωρήσουμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή, θα κροτηριάσουμε την ικανότητά μας ακόμα και στον εμπορικό αεροδιαστημικό τομέα, αλλά σίγουρα στο στρατιωτικό. Όλες αυτές λοιπόν οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει και μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη ε, εργατική δύναμη που δεν είναι μονάχα πολυάριθμη αλλά και σημαντική σε σχέση με τα προσόντα της. Αυτή η εργατική δύναμη υψηλά εξειδικευμένων εργαζομένων δεν μπορεί να διατηρηθεί άμα σταματήσουμε να έχουμε τα σχέδια ανάπτυξης. Θα χαθεί. Σκεφτείτε ότι έχουμε μια κυλιόμενη σκάλα η οποία κινείται συνέχεια. Ανεβαίνεται και μπορείτε να βγείτε ανα πάσα στιγμή. Αλλά όταν το κάνετε αυτό, συνεχίζει να γυρίζει η κυλιόμενη σκάλα. Άμα ξαναμπείτε, είσαστε σε μια άλλη θέση. Δεν είσαστε στην ίδια θέση που είσαστε. Υπάρχει αυτή η κυλιόμενη σκάλα της τεχνολογίας, όπου πρέπει να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας. <clears throat> Νομίζω λοιπόν ότι εδώ μπορώ να στραφώ και πάλι στον Ζωζ για να μας πει για τα επόμενα βήματα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, Ντέβιτ. Έχουμε αυτή τη στιγμή ε, τέσσερα βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της πρωτοπορίας της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας. Είναι τέσσερις βασικοί στόχοι λοιπόν και από τους οποίους θα πρέπει να απορρέουν αντίστοιχες δράσεις. Αν πιστέψουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις ικανότητες. Αυτές τις ικανότητες είναι φανερό ότι μπορούμε να τις εξασφαλίσουμε μόνο με συγκεκριμένα προγράμματα αναπτύξεως, ιδίως στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης για τις νέες τεχνολογίες. Και φυσικά αυτές θα οδηγήσουν εν καιρό σε ανάπτυξη πρωτοτύπων και παραγωγή. Δεύτερο σημείο, το οποίο ίσως δεν είναι τόσο προφανές, αναφέρθηκε προηγουμένως, Έχουμε τρία ευρωπαϊκά μαχητικά σε εξέλιξη ακόμα και σήμερα. Είναι σαφές όμως ότι αν είχαμε μια καλύτερη ορθολογικοποίηση ε, θα, δεν θα χρειαζόταν να έχουμε τρία αεροσκάφη αλλά ενδεχομένως και λιγότερα. Είναι σαφές ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να παραμείνουν στο στενοεθνικό χώρο. Καμία εθνική κυβέρνηση δεν έχει την επαρκή εθνική βιομηχανική βάση για να αναπτύξει τέτοια αεροσκάφη. Είναι πολύ ψηλές οι επενδύσεις και είναι μικρή η εθνική βιομηχανική δυνατότητα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα ευρωπαϊκό χώρο ανάπτυξης και κατασκευής αεροσκαφών μαχητικού χαρακτήρα. Επίσης, είναι αδιαφυσβήτητο και αυτό ισχύει και στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη, σε όλες τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες και οντότητες ότι για να μπορέσουμε <clears throat> να διατηρήσουμε αυτές τις ικανότητες η απόσταση μεταξύ της έναρξης ενός προγράμματος και της ε, συμπλήρωσής του που ανέρχεται σε 30 χρόνια περίπου ε, αυτή η απόσταση είναι μεγάλη ώστε να υπάρξει πάντα ο κίνδυνος για να χαθούν ε, ικανότητες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε και προγράμματα γεφύρωσης τα οποία θα εξασφαλίσουν θα διατηρηθούν αυτές οι ικανότητες όταν έχουμε να κάνουμε τόσο μακρά προγράμματα. Επίσης έχουμε ε, εντοπίσει και ορισμένα προγράμματα τεχνολογικής επίδειξης όχι μονάχα στον αεροδιαστημικό χώρο αλλά και στο έδαφος και εκεί στα προγράμματα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πάλι την ευρωπαϊκή ικανότητα. Εάν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες αυτές πρωτοβουλίες τότε όλες αυτές οι βιομηχανικές ικανότητες για την ανάπτυξη και την παραγωγή των στρατιωτικών αεροσκαφών και αυτό περιλαμβάνει και τα επαδρομένα και τα μη επαδρομένα αεροσκάφη θα χαθούν αυτές οι ικανότητες και θα είναι πολύ δύσκολο να επανακτηθούν και αυτό θα απαιτήσει πολύ χρόνο. Επομένως, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στις απαραίτητες δράσεις και θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον στρατηγό Μπρεβό. Ε, για να τελειώσουμε με τις ε, παρεμβάσεις, θα ήθελα να πω ότι η ανάλυση που έγινε από την Ακαδημία Αέρος και Διαστήματος και τα βασικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους συναδέλφους και από μένα σας επιτρέπουν να διαπιστώσετε ότι διατυπώνουμε μια σειρά από προτάσεις για να αποφύγουμε μια καταστροφική απώλεια της ικανότητας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σχολιάσω τις δύο πρώτες προτάσεις και να αναφερθώ στο γεγονός ότι καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε εκφράζοντας μια κοινή επιχειρησιακή ανάγκη. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι δεν θα πρέπει να αναμένουμε να τελειώσει η εργασία μας επί επιχειρησιακών θεμάτων και να περάσουμε στα τεχνολογικά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια κοινή έκφραση αυτής της ανάγκης. Από τη στιγμή που θα καθοριστεί αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μιλάμε για κάτι πολύ δύσκολο. Διαπιστώσαμε ε, ότι γίνονται συζητήσεις για να υπάρξει μια κοινή επιχειρησιακή ανάγκη οι συζητήσεις αυτές κατέληξαν κάπου, αλλά ε, με πολλές δυσκολίες. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος, θα πρέπει να πούμε ότι οι συζητήσεις αυτές ήταν πολύ δύσκολες. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ αναφέρθηκε ότι πριν να γίνει μια συζήτηση για τις κοινέ επιχειρησιακές ανάγκες θα πρέπει να ε, διεξαχθεί μια συζήτηση για το όραμα, για την προοπτική. Θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα έχουν τα πράγματα επιχειρησιακά τα επόμενα 20-30 χρόνια και μόνον μετά από αυτό θα μπορούσε κανείς να καταλήξει στον ορισμό μιας κοινή επιχειρησιακής ανάγκης. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια θαυμάσια αποστολή για την Ακαδημία. Αν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζητήσουν, οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας θα μπορούσαν να ε, βοηθήσουν τις ε, διάφορες χώρες για να αποκτήσουν μια κοινή προοπτική. Δεύτερο σημείο, ο Ευρωπαϊκός Φορέας χρηματοδότησε μια μελέτη σε όλες τις ευρωπαϊκές αεροβιομηχανίες που αναπτύσσουν δράσεις στον τομέα της άμυνας και ο τίτλος είναι Fast for Europe. Μία μελέτη πραγματικά αξιόλογη που προτείνει πραγματικά, πρακτικά μέτρα που θα επιτρέψουν την σύνταξη ενός οδικού χάρτη για τα μαχητικά αεροσκάφη. Και μεταξύ των πρώτων στοιχείων αυτού του οδικού χάρτη διαπιστώνουμε ότι το πρώτο είναι να διασωθεί η τεχνολογία. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα θα χαθεί αυτός ο τομέας. Μιλάμε ιδιαίτερα στον, ε, για την τεχνολογία στον τομέα της ηλεκτρονικής. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε, δεν μιλάμε για ιδιαίτερα δαπανηρές ε, δράσεις, καμία σχέση με τα δισεκατομμύρια που δίνονται για άλλα προγράμματα. Αυτή η ε, ικανότητα θα διατηρηθεί μόνο με προγράμματα εξυγχρονισμού που αφορούν και τον επιχειρησιακό τομέα που χρειάζεται να, αναπτύσσει, ε, να αναβαθμίζει το υλικό του αλλά και τη βιομηχανία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στο συνάδελφο Ζορτ Μπιντέλ για να συνεχίσει για τα πέντε άλλα σημεία. Καταρχήν επιτρέψτε μου να πω κάτι σχετικά με την βιομηχανική συνεργασία. Κοιτάξτε, δικό μας καθήκον δεν είναι να χαράσουμε βιομηχανική πολιτική. Εμείς ε, το πολύ πολύ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρουσιάζουμε τα γεγονότα και να καταδεικνύουμε ίσως ε, κάποιες ε, συνέπειες. Αλλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε στα οργανωτικά. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία σταθεροποιηθεί, κυρίως σε αυτό τον τομέα, στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, προγραμμάτων επίδειξης, αυτό θα είναι επικοδομητικό. Γιατί υπάρχουν πολλές ε, βιομηχανικές δυνατότητες που αναπτύσσονται παράλληλα και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξοικονομήσουμε δαπάνες. Έχοντας κατά νου αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα κλασικά μοντέλα συνεργασίας, να αναζητήσουμε νέες μορφές συνεργασίες στο βιομηχανικό τομέα, ας πούμε, παραδείγματο χάρη, να υπάρχει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική δομή ε, για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ε, για ένα πρόγραμμα επίδειξης ε, ε για τα μαχητικά αεροσκάφη αυτά αποτελούν μόνο ένα τμήμα των δυνατοτήτων που μπορούμε να αναπτύξουμε. Η εμπειρία βέβαια μας έχει αποδείξει ότι όλες οι δυνατότητες βιομηχανικής σταθεροποίησης αποτυγχάνουν κατά κανόνα αν η τάση αυτή δεν βασίζεται σε ένα πρόγραμμα demonstrator ή σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς ε, να περιμένει από τη βιομηχανία να συνενώσει τις δυνάμεις της ε, για ένα θέμα όπου δεν υπάρχει καμία προοπτική. Και εξ αυτού απορρέει το ότι σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο άμυνας πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις για προγράμματα που δεν αποτελούν αυτό σκοπό αλλά έχουν ως στόχο να καλύπτουν ανάγκες. Και αυτό μόνο ως παρατήρηση αλλά νομίζω ότι είναι και αυτονόητο αυτό που σας είπα. Τώρα θα δώσω το λόγο ε, στο συνάδελφο David Marshall ο οποίος θα ολοκληρώσει και αυτή την παρέμβασή μας. Ευχαριστώ Τζος, και πάλι. Εν συμπεράσματι θα ήθελα να κάνω τα εξή σχόλια. Υπάρχει ένα μεγάλο ιστορικό πολυεθνικών προγραμμάτων στον αμυντικό τομέα και βέβαια δεν είχε πάντα την μεγαλύτερη δημοσιότητα. Δεν είχαν πάντα τη μεγαλύτερη δημοσιότητα γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να φτιάξει κανεί ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο θα ικανοποιήσει όλου. Και για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να δεχτούν όλοι συμβιβασμού. Ξέρουμε όμως ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γιατί υπήρξαν τέτοια επιτυχημένα προγράμματα και φυσικά στον εμπορικό τομέα είναι το πιο ε, επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας στην Ευρώπη, το consortium του Airbus που έδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί στον τομέα αυτό. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο σε στρατιωτικό επίπεδο με ένα μικρό αριθμό εθνών που είναι έτοιμα να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία αλλά που θα είναι ανοιχτό και σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη να συμμετάσχουν, εφόσον φυσικά η συμμετοχή τους δεν μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα του προϊόντος, γιατί αλλιώς αρχίζει να μειώνεται η αξία ενός τέτοιου εγχείρηματο. Το πρώτο όμως απαιτούμενο το οποίο χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια τέτοια συνολική ενέργεια είναι κατά την άποψή μου μια δήλωση πολιτικής θέλησης, ότι η Ευρώπη θέλει πράγματι να έχει κάτι τέτοιο. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεκινήσει. Όλο, όλο αυτό πρέπει να ξεκινήσει με ένα αρχέτυπο, με ένα μοντέλο επίδειξης το οποίο θα οδηγήσει εν καιρό στο τελικό προϊόν. Όπως ακούσατε υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη τεχνολογίας και αυτό θα δώσει ωφέλη τα οποία θα κατανεμηθούν με πιο ευρύ τρόπο στη συνέχεια στη βιομηχανία. Όλα αυτά, όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα μακροχρόνιο και καλά ζυγισμένο σχέδιο επένδυσης. Δεν σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να πούν οι χώρε ότι θα πρέπει να καταβάλουν κάποια ποσά, αλλά θα πρέπει να ξέρουν πω ποια κατεύθυνση κινούνται. Αυτή η πολιτική θέληση λοιπόν δημιούργησε την επιτυχία του Airbus. Χρειαζόμαστε την αντίστοιχη πολιτική θέληση για να υπάρξει ένα επιτυχημένο, μια επιτυχημένη βιομηχανία μαχητικών αεροσκαφών. Ελπίζω ότι σας έχουμε πείσει γιατί χρειαζόμαστε πράγματι μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στα θέματα αυτά. Απλώς ένα σύντομο σχόλιο πρωτού δώσω το λόγο στην συζήτηση και την ανταλλαγή ερωτημάτων και απαντήσεων. Πιστεύω ότι καταλάβατε με, τα, με την παρέμβαση και μου του ιδίου και των δύο συναδέλφων μου ότι πράγματι χρειάζεται μια υποστήριξη της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας η οποία είναι αξιοσημείωτη και υποστηρίζει την ελληνική πολεμική αεροπορία η οποία είναι και αυτή εξαιρετική και πάρα πολύ αποδοτική. Βλέπετε ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου γίνονται λίγες ενέργειες και υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί αυτή η ικανότητα. Εμείς έχουμε υποβάλει ήδη μια σειρά από προτάσεις που σας παρουσιάσαμε προηγουμένως. Μπορούν να υπάρξουν και άλλες προτάσεις, αλλά σίγουρα το βασικό είναι φανερό ότι είναι να υπάρξει πολιτική θέληση. Αυτό που θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει είναι να υπάρξει μια κινητοποίηση για το ζήτημα αυτό και οι λήπτες αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και να προχωρήσουν σε δύο είδη δράσεων. Μια πρώτη δράση θα πρέπει να είναι να υπάρξει μεγαλύτερη κίνηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, η οποία μπορεί να δουλέψει μονάχα με αίτηση των κρατών μελών και να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας να προχωρήσει σε έρευνα των δυνατοτήτων και των απαραίτητων προϊόντων που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να δημιουργήσει το οδηγό νήμα το οποίο <clears throat> θα οδηγήσει στην τεχνολογική ανάπτυξη, στα, στα προϊόντα επίδειξης και μετά στα ε, μαχητικά αεροσκάφη και την κατασκευή τους. Αυτό λοιπόν απαιτεί δράση των κρατών μελών και η δεύτερη δράση την οποία θα θέλαμε να δούμε είναι να υπάρξει κάποια κίνηση από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 και θα θέλαμε να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τα προβλήματα αυτά που μπορεί να οδηγήσει στην ε, πολιτική θέληση να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε τις ερωτήσεις των κυρίων κοινοβουλευτικών. Σας ευχαριστώ πολύ, Λέω Πρόεδρος. Πιστεύω ότι ήταν ε, πάρα πολύ σαφής η παρέμβασή σας. Μάθαμε πάρα πολλά ενώ παράλληλα η παρέμβαση είχε πάρα πολλές πολιτικές χρειές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να στραφούμε σε ένα παράδοξο. Γιατί παρόλο που ο τόνος της εισαγωγικής παρέμβασης ήταν μάλλον αρνητικό αφού αναφερόμασταν στο η πιθανότητα μείωσης της ικανότητας στην Ευρώπη, όταν κοιτάμε την κατάσταση διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα αφορά το υπερβολικό, το πλεόνασμα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που αναπτύσσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική στον τομέα των εξαγωγών. Δεν βλέπουμε αυτή την πτωτική τάση, μάλλον βλέπουμε μια ανωδική πορεία, μια ε, υπερβολή. Βεβαίως μιλάμε για προθεσμίες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την έρευνα. την ε, χρήση ορισμένων μέσων. Βρισκόμαστε πάρα πολύ μπροστά και βεβαίως αυτή η προοπτική είναι που μας προβληματίζει στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε αυτή την υπενθύμηση. Επίσης είναι χρήσιμο αλλά και ευχάριστο να αναφέρω για μία ακόμα φορά μιλώντας για ένα τομέα βιομηχανικό, ένα τομέα που αφορά τις ικανότητες, ότι όλα θα εξαρτηθούν από το στρατηγικό πλαίσιο που θα οριστεί εκ των προτέρων. Και στην Ευρώπη στο Συμβούλιο Κορυφής δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομίες όταν μιλάμε για θέματα στα οποία θα πρέπει να συμπορευτούμε στον τομέα της αμυντικής πολιτικής. Το να αποφασίσουμε να αποκτήσουμε ικανότητες χωρίς να γνωρίζουμε σε τι πλαίσιο θα κινηθούμε τα επόμενα 20-30 χρόνια δεν έχει και πολύ νόημα. Η στρατηγική συζήτηση λοιπόν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν <clears throat> την ικανότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι αυτονόητο, αλλά δεν βρίσκει σύμφωνους πολλούς από τους συνομιλητές μας στα πλαίσια του Συμβουλίου, όπου πολλοί πιστεύουν ή κάνουν ότι πιστεύουν ότι θα αρκεστούν μερικές ανακοινώσεις για την κοινή ικανότητα για να υπάρξει μια πραγματική προσπάθεια στον τομέα της άμυνας. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Από αυτή την άποψη, συνεπώς, Καταλαβαίνω τις δικές σας προσδοκίες που ταυτίζονται με τις δικές μας, ότι δεν πιστεύω ότι το Συμβούλιο αυτό καθ' αυτό θα μπορέσει να πάρει αποφάσεις καλά δομημένες. Τουλάχιστον ελπίζουμε να μπορέσουν το σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Το δικό μου ερώτημα, συγκεκριμένο ερώτημα, <clears throat> αφορά την ανακοίνωση που έγινε για τα αεροσκάφη χωρίς ε, χειριστή κατά τη διάρκεια του σαλονιού του Μπουρζέ από τρεις κατασκευιστές σε ό,τι αφορά την διάθεσή τους για να κατασκευάσουν ένα ευρωπαϊκό σκάφος ε, ε, τηλεχειρισμού. Εσείς τι πιστεύετε, νομίζετε ότι διαφαίνεται κάτι ε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι σε επίπεδο αεροσκαφών χωρίς ε, χειριστές από αυτές τις επιχειρήσεις αλλά και από άλλους. Αυτό το είδος της ανακοίνωσης, αυτό το είδος του προγράμματος θα μπορούσε να αποτελεί προάγγελο κάποιου άλλου πράγματος ε, για τα ε, αεροσκάφη με χειριστή ή θα παραμείνουμε σε αυτό το στάδιο έρευνας ε, για τα αεροσκάφη χωρίς χειριστή. Ο κύριος Πάσκου. Well, thank you very much. I... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω μετά από το φόρουμ των Παρισίων. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω για την τόσο σημαντική αυτή συνάντηση. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την παρέμβασή σας. Γιατί είναι αυτό που μας χρειαζόταν για να μπορέσουμε να καθορίσουμε σαφώς τις προτεραιότητές μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ενδεχομένως ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα διαμορφώσει τις ανάγκες μας το μέλλον θα είναι οι αποστολές CSDP και δεύτερον αυτό που βρίσκεται πάντοτε στη βάση, η ικανότητα της Ευρώπης να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Νομίζω ότι ξέρετε ότι από τη στιγμή που θα αρχίσετε να σκέφτεστε το θέμα της εξαγωγής των αεροσκαφών, ε, αυτό βεβαίως είναι μια ξεχωριστή ιστορία, αλλά πιστεύω οι αποστολές του CFD, ε, CSDT, του ΣΚΕΠΑ δηλαδή, θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Κανένας βεβαίως δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής διαπαντός ότι από τη στιγμή που θα φτάσει αυτό το επίπεδο δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με κινδύνους. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχουν δύο τάσεις που είναι ορατές. Η μία φορά την βιομηχανία και τον στρατιωτικό τομέα. Και οι δύο αυτοί τομεί επικαλύπτονται ως ένα βαθμό γιατί ξέρετε ότι υπάρχει τάση για ανάληψη πολλαπρών ρόλων. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί. Έχουμε αεροσκάφη που είναι ικανά να διεισδύουν ε, σε υψηλό ή χαμηλό επίπεδο άμυνας Όλα αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα αεροσκάφος και μόνο. Και πιστεύω ότι αυτός ο πολλαπλός ρόλος θα συνεχιστεί. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει ένα συνδυασμός με τα αεροσκάφη χωρίς χειριστή που θα πρέπει να ακολουθήσουν τη δική τους ανεξάρτητη πορεία. <clears throat> Το δεύτερο, ξέρετε ότι ο στρατιωτικός τομέας για να μπορέσει να επιβιώσει και για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το χώρο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει ένα θύλακο μέσα στην, ε, ε, ε, ε, στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι ο ένας τομέας. Ξέρετε ότι υπάρχουν τα χρήματα γενικά για την έρευνα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα χώρο για τον τομέα της άμυνας. Μιλάμε βεβαίως για την ενιαία αγορά. Και αν ρίξετε μια ματάκια στον ουρανό βλέπετε και τον ενιαίο ουρανό. Εδώ θα πρέπει να ενσωματώσουμε, να εντάξουμε τα αεροσκάφη χωριστηρίκηστη, τα στρατιωτικά αεροσκάφη κτλ. Αυτή είναι μια δεύτερη ε, στάση, <clears throat> δηλαδή ε, συμπόρευση της πολιτικής και της πολεμικής αεροπορίας. Να δούμε πώς θα μπορούσε να ενσωματωθεί, να ενσωματωθούν τα στρατιωτικά αεροσκάφη στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Είπατε ότι <clears throat> χρειαζόμαστε κάποια ελαστικότητα στον τομέα το βιομηχανικό για να μπορέσουμε άμεσα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Αλλά χρειαζόμαστε μια βιομηχανία η οποία ε, δεν έχει αφυπνιστεί ακόμα. Χρειαζόμαστε μια ακμαία βιομηχανία η οποία παράγει και μπορεί να διατηρεί την ελαστικότητά της. Θα έλεγα ως προς το Συμβούλιο, τον Δεκέμβριο του τελευταίου Συμβούλιο που τα συζήτησε τα θέματα αυτά ήταν το 2008, στην αρχή της κρίσης. Πολλά πράγματα έχουν συσσωρευτεί στο μεταξύ και βεβαίως δεν θα πρόκειται για θετικά. Αντίθετο, θα έλεγα ότι παρατηρήθηκε μια υποβάθμιση σε πολλούς τομείς ως προς την ευρωπαϊκή άμυνα. Ενδεχομένω περιμέναμε πάρα πολλά από αυτό το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο αυτό θα υιοθετήσει βασικές αποφάσεις που θα διανοίξουν ε, δρόμους και βεβαίως ότι θα υπάρξει ένα σύστημα παρακολούθησης. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο πιστεύω ότι υπάρχουν δύο σημαντικές ανάγκες. Καταρχάς θα υπάρξει ένα είδος moratorium έτσι ώστε οι χώρες να σταματήσουν, τα κράτη να σταματήσουν να μειώνουν τους προϋπολογισμούς για την άμυνα. Ένα moratorium, οποιαδήποτε μορφή και να προσλάβει. Και δεύτερον, αυτή είναι μια ιδέα που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ενδεχομένως ε, χρειαζόμαστε μια πολιτική δήλωση ως προς το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Γιατί σκεφτείτε ότι η Ευρώπη θέλει να είναι ένα σημαντικός διεθνής φορέας. Για να μπορέσει να το καταφέρει θα πρέπει να διατηρηθεί η τεχνολογική ικανότητα. Την έχουμε, αλλά ε, υπάρχει κίνδυνος να τη χάσουμε. Αν θέλετε να διατηρηθεί η ε, τεχνολογία, εμείς θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, Ξέρετε ότι αυτού του είδους τα πράγματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε τέτοιου είδους πολιτικές δηλώσεις, γενικές πολιτικές δηλώσεις του Συμβουλίου. Και από τη στιγμή που το Συμβούλιο θα χαράξει αυτές τις στρατηγικές γραμμές, αφού είμαστε πεπισμένοι θα ζητήσουμε στις χώρες μέλη να συμμορφωθούν και θα περάσουμε στην επόμενη φάση που είναι το moratorium. Ε, προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το 2% του ε, ΑΕΠ και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και εδώ. Έχω απόλυτη συνείδηση ότι θέλετε να μας κάνετε να συνειδητοποιήσουμε τις ευαισθησίες και ε, τα προβλήματα της βιομηχανίας. Βεβαίως θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των αποφάσεων το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ κύριο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την υποεπίτροπή μας. Κατανοώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση με τη βοήθεια των προτάσεων που μας παρουσιάσατε. Πολλά θέματα μπορεί να είναι αμφιλεγόμενα, αλλά σίγουρα η κατάσταση έχει, ε, έχει γίνει πιο έντονη και πιο δύσκολη λόγω των τελευταίων εξελίξεων και πρέπει τελικά να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα και να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ έχω ήδη ο ίδιος αντιμετωπίσει προσωπικά τα θέματα αυτά στη χώρα μου των μαχητικών αεροσκαφών και επομένως γνωρίζω την προβληματική την οποία παρουσιάσατε και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα Υπουργεία Άμυνας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι είναι σοβαρά μέλη του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι και η Πολωνία, η χώρα μου. Και είμαστε μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι αμυντικοί προπολογισμοί δεν μειώνονται. Τουλάχιστον 2% του προϋπολογισμού μας πηγαίνουν στην άμυνα και ένα μεγάλο μέρος από αυτά πηγαίνει για τον εξυγχρονισμό της αεροπορικής ε, ε, βιομηχανίας και θέλουμε να περάσουμε από τα Σούχοϊ και τα ΜΙΚ στη δυτική τεχνολογία μαχητικών αεροσκαφών. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζει και η υποεπιτροπή μας ότι όλες οι στρατιωτικές συγκρούσεις αποφασίζονται τελικά στον αέρα. Δεν μπορεί κανείς να επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους χωρίς αεροπορική υπεροχή. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό πρόβλημα. <clears throat> ένα δεύτερο θέμα είναι ότι η στρατιωτική τεχνική, ιδίως αυτή στην η αεροπορική τεχνική είναι ιδιαίτερα πολυδάπανη και πολύπλοκη και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο μπορεί να κοστίζει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος. Και ένα τρίτο πρόβλημα που θέλω να επισημάνω θα πρέπει να έχουμε όλο και μεγαλύτερη προσοχή στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα οποία, και αυτό είναι ε, απόλυτα σωστό να γνωρίζουμε ότι η ικανότητα στον τομέα αυτό των μη επανδρομένων αεροπλάνων είναι σημαντική. Τα, θέματα, τα μη επανδρομένα αεροπλάνα μας βοηθούν να αποφύγουμε την απώλεια ανθρωπίνων ζώων, λέει ο μιλητής. Και είπε και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ντανζάν, ότι έχουμε ένα βασικό ερώτημα να απαντήσουμε. Το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις δικές της ικανότητες, τις αυτόνομες της ικανότητες στον τομέα της χρήσης των στρατιωτικών αεροσκαφών και αν θέλει να αναπτύξει την αντίστοιχη τεχνική. Είναι προφανώς πολύπλοκη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί για τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αναφέρομαι εδώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στις χώρες του ΝΑΤΟ είναι φανερό ότι θέλουμε να έχουμε δυνάμεις στρατιωτικές οι οποίες είναι συμβατές με το ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό θέλουμε να δούμε, είναι σημαντικό να απαντήσουμε το ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να λειτουργήσει αυτόνομα από το ΝΑΤΟ και να δημιουργήσει ιδιαίτερες στρατηγικές και αναπτύξεις αεροσκαφών ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο ΝΑΤΟ. Είδαμε στην Λιβύη και στο Μάλι πώς, πόσο σημαντική είναι μια ευρωπαϊκή αεροπορία. Αλλά θα είπατε αυτά κάπως ευγενικά και δεν αναφέρατε ότι χωρίς την αμερικανική υποστήριξη δεν θα μπορούσαν να έχουν λάβει χώρα καν αυτές οι στρατιωτικές επιχείρησεις. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω μερικά περαιτέρω στοιχεία της προβληματικής. Τα μαχητικά αεροσκάφη της πέμπτης γενιάς είναι το πρώτο θέμα. Θα πρέπει εμείς να συνασπιστούμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι ίσως βρίσκονται στον δρόμο για να το κάνουν αυτό. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο. Εγώ νομίζω δεν έχουμε καμία εναλλακτική λύση και δεν μπορούμε να μην το πράξουμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε. Εμείς θα πρέπει να έχουμε και μια κοινή αντίληψη σε σχέση με τα μαχητικά αεροπλάνα. Εγώ έχω πετάξει με το F-16, το Eurofighter, το Griffon, το, τα Mirage. Γνωρίζω αυτά τα αεροσκάφη, τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη είναι περισσότερο πλατφόρμες για αναγνωριστικά συστήματα και οπλικά συστήματα. Αν συζητάμε για τα νέα αυτά αεροσκάφη, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση και στα μέσα αναγνώρισης αλλά και στα οπλικά συστήματα που φέρουν αυτά τα αεροσκάφη και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο πρόβλημα τα προγράμματα ανάπτυξης αυτών των οπλικών συστημάτων και των συστημάτων αναγνώρισης είναι ιδιαίτερα πολυδάπανα συστήματα και απαιτούν μια ικανότητα να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτά τα θέματα τα οποία τονίστηκαν ορθά από τον πρόεδρό μας και είναι η απάντηση του αν θέλουμε μια ικανότητα στον ευρωπαϊκό χώρο για αυτά τα συστήματα και η απάντηση δική μου είναι ναι. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Μια διευκρίνηση μονάχα σε ό,τι αφορά την συνάρθρωση των ενεργειών μας με αυτές των Αμερικανών. Η υποστήριξη των Αμερικανών στη Λιβύη και, στη, και στο Μαλί είναι αποφασιστική βέβαια η υποστήριξη των Αμερικανών, αλλά όπως είπαν και οι ομιλητές μας, από την ε, πλευρά της Ευρώπης υπάρχει η αυτόνομη δυνατότητα να εισέλθουμε σε ένα θέατρο μάχης. Τα Ραφάλ, τα οποία το Μάρτιο πέταξαν πάνω από την, ε, το Μάρτιο 2011 πάνω από τη Βενγάζη, το κάναν χωρίς εξωτερική υποστήριξη, <clears throat> είτε σε ό,τι αφορά την ε, επίθεση κατά των αντιαεροπορικών εγκαταστάσεων της ε, Λιβύης, είτε σε ό,τι αφορά την, τον ανεφοδιασμό τους, δεν χρειάστηκαν καμία υποστήριξη από τους Αμερικανούς. Επομένως, οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε μια τέτοια πολεμική ενέργεια ε, αυτόνομα, χωρίς να χρειάζονται την υποστήριξη των Αμερικανών για ανεφοδιασμό ή συλλογή πληροφοριών. Αυτό είναι λοιπόν μια ε, διευκρίνηση που ήθελα να κάνω. Ο Ανδρέας Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό στον κύριο Πάσκο, θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από τα κράτη-μέλη να πάψουν να περιορίζουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς ε, υπό τις παρούσες συνθήκες. Ίσως πουν ότι θα το κάνουν, αλλά δεν θα το κάνουν. Αν καταλαβαίνετε βέβαια τι εννοώ. Ελπίζω να μπορεί κανείς να αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμόσει οικονομίες κλίμακος, σχέση κόστους ωφέλους, βελτιωμένες τεχνολογίες και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει. Για να μπορέσει λοιπόν η βιομηχανία να παρουσιάσει ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια νέα γενιά μαχητικών αεροσκαφών και για να μπορέσει να αποδείξει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, υποχρησιμοποιείται, αυτό είναι ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε καλύτερα. και πρέπει να αναζητήσουμε την καλύτερη δυνατή προσέγγιση ε, για να δούμε ε, πώς ε, για να δούμε πώς μπορούμε να προβάλλουμε τα επιχείρηματά μας που θα πείσουν τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Κοιτάξτε, πρέπει να ληφθούν ε, σοβαρές ε, αποφάσεις σχετικά ε, με τις προμήθειες και τη χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, την καλύτερη χρήση. Αυτό θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ε, εγκρίνετε οι αμυντικές προμήθειες να ενταχθούν στις διαπραγματεύσεις ή μήπως διαφωνείτε με αυτό. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο βέβαια οδηγεί και σε διχογνωμίες μεταξύ μας. Έχετε το λόγο λοιπόν να απαντήσετε εφόσον επιθυμείτε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θέσατε τόσο σημαντικά αυτά τα ερωτήματα. Εγώ θα καταβάλω μια προσπάθεια να διευκρινίσω ορισμένα σημεία τα οποία τα κατέχω και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου για να αναφερθούν σε άλλα σημεία που είναι δική τους αρμοδιότητας. Καταρχάς ετέθη ερώτημα σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση για τα αεροσκάφη χωρίς ε, ε, χειριστή αναγνώρισης, ε, αναγνώριση θα ήθελα να κάνω μια πρώτη παρατήρηση, τα αναγνωριστικά με συγχωρείτε αεροσκάφη. Σε ό,τι αφορά το θέμα αναγνωριστικών ε, αεροσκαφών ε, και αεροσκαφών παρατήρησης, όλοι λένε ότι μπορούν να παράγουν τα πάντα. Τίποτα όμως ε, δεν προχωράει στην Ευρώπη, ενώ τα πράγματα εξελίσσονται από πλευράς Αμερικανών. Σας το λέω γιατί αυτό διαφέρει κάπως από τα, σε σχέση με τα μαχητικά αεροσκάφη και τα αεροσκάφη δίχως χειριστή. Το ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό μας δείχνει το τι θα πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση των μαχητικών. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με τρεις χώρες που προσπαθούν να το κάνουν με βάση επίσημες αποφάσεις που προσπαθούν λοιπόν να κάνουν τον πυρήνα ενός προγράμματος το οποίο μετά θα το παραλάβουν άλλοι. Υπάρχουν λοιπόν δύο-τρεις ε, χώρες ε, οι οποίες ε, πραγματικά ορίζουν έναν ανάδοχο που θα αναλάβει να εξελίξει αυτό το πρόγραμμα. Στον τομέα αυτό λοιπόν των αεροσκαφών χωρίς χειριστή διαπιστώνουμε ότι καταβάλλεται μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πασκού για την παρέμβασή του. Ο κύριος Πασκού είπε πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη το θέμα της άμυνάς της. Βεβαίως είναι ένα θέμα πολύ μεγάλης σημασίας για σας που εκπροσωπείτε τους λαούς της Ευρώπης. Παρατήρησα κάτι. Η Ευρώπη είτε με το ΝΑΤΟ είτε μόνη της συμμετείχε στην ε, ε, πρόσφατες σειράξεις και θα ήθελα να πω ότι τα σκάφη που σχεδιάζονται και που απεδείχθη ότι είναι αποτελεσματικά είναι τα ίδια που εξασφαλίζουν την ασφάλειά μας, είναι τα ίδια που έχουν τον ίδιο εξοπλισμό, την ίδια αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να αναφερθώ, να αναφέρω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν αρχίζει στα σύνορά της. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει το θέμα της γυτνίασης. Εμείς είμαστε ο κήπος της Ευρώπης που λαμβάνουμε πάρα πολλές απειλές και δυνητικές απειλές. Η απειλή μας προσεγγίζει και με την, στην περίπτωση του Μαλή και της Λιβύης η απογείωση των αεροσκαφών έγινε από την Ευρώπη. Προσεγγίζει λοιπόν η απειλή και εδώ ακριβώς μπορούμε να κατανοήσουμε το ρόλο της ε, προάσπισης της Ευρώπης, της άμυνας στην Ευρώπη. Έγιναν παρατηρήσεις και για θέματα εξαγωγών. Εξαγωγές, γιατί το καταλαβαίνετε κι εσείς, οι εξαγωγές είναι ένας τομέας ιδιαίτερα σημαντικός σε επίπεδο στρατηγικό, ε, σε επίπεδο ε, ρόλου στην Ευρώπη. Αλλά για να γίνουν εξαγωγές θα πρέπει να υπάρχει ένα προϊόν εξαγωγών. Για, αν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε, χάνουμε την επιρροή μας ε, στην Ευρώπη και αυτό πραγματικά θα αποβεί καταστροφικό. Αναφέρθηκε και η σημασία του πολλαπλού ρόλου και τις ικανότητες ε, και των ικανοτήτων μπορούμε να έχουμε εκεί. Διαπιστώσαμε, το διαπιστώσαμε αυτό στη σύγκρουση στο Μαλί. Τα αεροσκάφη ε, εκεί μπορούσαν στην ίδια ε, αποστολή να εκτελέσουν πολλές ε, λειτουργίες περνώντας από την, ε, να εκτελέσουν πολλές λειτουργίες περνώντας από τη μία στην άλλη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση για τα μελλοντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο συνδυασμός, η συνεργασία με την πολιτική βιομηχανία επίσης είναι σημαντικός στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς των νέου ουρανού. Είναι βεβαίως ε, σαφές ότι υπάρχουν σημαντικές ε, ε, σχέσεις που αναφέρθηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα το θέμα της πτήσης αεροσκαφών χωρίς χειριστή στον πολιτικό αέριο χώρο που είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαφές ότι υπάρχει μία δραστηριότητα μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών δράσεων. Δεν θα απαντήσω βεβαίω σε όλα τα θέματα. Να αναφερθώ στον κύριο Ζέμκε. Ο κύριος Ζέμπκε είπε ότι η Πολωνία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ως προς αυτό το θέμα. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το πρόβλημα των μαχητικών αεροσκαφών δεν αφορά μόνο τις έξι χώρες, αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο τομέας που καλύπτεται από τα αεροσκάφη αυτά είναι ευρύτατος, αφορά πολλές πτυχές τεχνολογίας. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, ευρωπαϊκές ε, χώρες ε, που ενδιαφέρονται και δεν θα πρέπει να φοβούνται να πάρουν μέρος σε μεγάλα προγράμματα μέσα από με διάφορους τρόπους και οι χώρες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να εκφράσουν την επιθυμία τους ναι, για συμμετοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις δικές της δυνάμεις. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της κοινή ασφάλειας που εξασφαλίζεται από το ΝΑΤΟ. Κοινή ασφάλεια. Επαναλαμβάνω, κοινή. Ο, το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν μια ομπρέλα ή μια διασφάλιση. Αποτελεί ένα σύνολο χωρών, μια ομάδα χωρών και το, το ΝΑΤΟ είναι τόσο ισχυρό όσο είναι οι χώρες που το ε, απαρτίζουν. Ξέρετε για το 50% που πρόσφατα αναφέρθηκε. Σε ό,τι αφορά το 50% θα πρέπει να εξασφαλιστεί και με αποτελεσματικότητα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Όταν ήμουν υπεύθυνο για στον τομέα των επιχειρήσεων, παρατήρησε ότι οι Αμερικανοί θα ήθελαν να αποσυρθούν. Δεν ήθελαν να πάρουν μέρος σε δράσεις που ξεκινούσαν από ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι μου έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν, δεν θα γίνει ποτέ. Και όμως έγινε δύο φορές με τη Λιβύη και με το Μάλι. Στη Λιβύη είναι χαρακτηριστικό, γιατί ξεκίνησαν και μετά αποχώρησαν από τις επιχειρήσεις. Βεβαίως, είναι αλήθεια, είναι πολύ σημαντική η αποστήριξη σε περιπτώσεις που δεν ε, αρκούμε στην Ευρώπη, αλλά δείξαμε την ε, ικανότητα που έχουμε στην Ευρώπη, όπως το τόνισε εξάλλου και ο κύριος Πρόεδρος. Également un euh, Άλλο τομέα που συνδέεται με το ΝΑΤΟ <clears throat> και το θέμα των προτύπων. Δεν ε, έχουμε απόλυτη συνείδηση αυτού το γεγονός ότι η Ευρώπη αναπτύσσει μια μαχητική βιομηχανία σημαίνει ότι η Ευρώπη θα είναι ισχυρή για να επιβάλλει τα δικά της τα πρότυπα και να τα ορίσει τα πρότυπα. Τι συμβαίνει τώρα, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εκείνε που ορίζουν τα πρότυπα και τα επιβάλλουν στο ε, ΝΑΤΟ. Και βεβαίως κανείς δεν αντιτίθεται σε αυτό. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ότι ε, επιβάλλουν αυτά τα πρότυπα στους άλλους. Η Ευρώπη αναπτύσσοντας τα δικά της πρότυπα θα μπορούσε να φύγει από αυτή τη θέση εξάρτησης. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλλα σημεία και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Αναφέρθηκε ότι ότι ο Ευρωπαϊκός Φορές Άμυνας ε, δεν χρησιμοποιείται με παραδειγματικό ε, τρόπο όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες αποστολές για, αυτή την, ε, για αυτό και αυτόν τον οργανισμό. Βεβαίως ο προϋπολογισμός της είναι ανεπαρκής και χρειάζεται περισσότερα κονδύλια. Βεβαίως, πριν να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να αναλάβει μία αποστολή, η οποία δεν είναι δαπανηρή, και αφορά τον ορισμό μιας κοινή πρόπτικης, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια θαυμάσια αποστολή που θα επιτρέψει στην ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα να πτύξει τον ρόλο του. Αυτό θα μπορούσε να διαδραματίσει τον ρόλο του. Αυτό θα μπορούσε να γίνει το 2013. Τώρα, αν συμφωνούμε για τις διαπραγματεύσεις ε, που γίνονται ε, στον τομέα της ε, άμυνας. Βεβαίω υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ενδεχομένω οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να επεκταθούν ω προ αυτό το θέμα. Να σα δώσω το λόγο. Δεν ξέρω ποιο θέλει να μιλήσει πρώτο. Απελθέτω απ' εμού. Ευχαριστώ. Ένα-δύο σημεία μονάχα θέλω να αντιμετωπίσω κυρίω από τον κύριο Πάσκου. Ένα κομβικό θέμα όπως αναφέρατε είναι το θέμα του πώς στην Ευρώπη μπορούμε να ενσωματώσουμε καλύτερα αυτά τα οποία δαπανούμε στην ε, πολιτική αεροπορία και αυτά τα οποία δαπανούμε για την πολιτική, πολεμική αεροπορία. Στον ε, τομέα της πολιτικής αεροπορίας υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προτείνει η βιομηχανία μαζί με την Κομισιόν για την υποστήριξη αυτή και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άμεση σχέση με τις ανάγκες στον αμυντικό τομέα. Και δεν βλέπω γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι σαν να έχετε μια εταιρεία που λέτε έχω κάποια στρατιωτικά προϊόντα, κάποια πολιτικά προϊόντα, αλλά οι δύο, τα δύο τμήματα της επιχείρησης δεν έχουν καμιά επαφή μεταξύ τους. Εγώ νομίζω μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή η κατάσταση. Και αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Νταφ. Έχει δίκιο. Δεν θα υπάρχουν ε, οι δυνατότητε σε οικονομικό επίπεδο. Θα ήταν χρήσιμο όλοι να δαπανούν το 2% του ΑΕΠ τους, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτό. Ο μόνος άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μπορεί να γίνει αυτό καλύτερα με μια καλύτερη ε, συνεργασία του πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, αλλά και με καλύτερη ε, συνένωση των πελατών μας, γιατί ο κατακαιρματισμός δεν μας βοηθάει. Λοιπόν, η συνένωση και σε επίπεδο βιομηχανικό και σε επίπεδο πελατών θα πρέπει να γίνει προς όφελος της αποδοτικότητας. Αν υπάρξει λοιπόν μια πολιτική δήλωση το Δεκέμβριο, θα μπορούσε να κινητοποιήσει όλους. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη βιομηχανία που λέει μπορούμε να κάνουμε πράγματα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πράγματα, αλλά γιατί και πώς θα επενδύσουμε και θα πούμε στους μετόχους μας ότι είναι καλή επένδυση εάν δεν έχουμε καθόλου κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι οι πελάτες μας θέλουν και αυτοί να υπάρξει επένδυση και ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτή. Και για τις ΗΠΑ, τώρα μιλάω για σε εμπορικό επίπεδο, δεν είμαι γνώστης των λεπτομεριών για την εμπορική συμφωνία. Αλλά ουσιαστικά βασίζονται στην έννοια της αμφιδρομίας, ότι τα πράγματα θα πρέπει να βασίζονται σε κάποια μορφή αμοιβαιότητα, σε κάποια μορφή μια συμφωνίας που είναι αμοιβαίως επωφελή. Αυτό το λέμε στα αγγλικά, στα βρετανικά, ότι θέλουμε να έχουμε ένα γήπεδο που είναι ισόπεδο. Αλλά δεν είναι παιχνίδι, δεν μιλάμε για γήπεδο σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό που πιστεύω θα θέλανε να έχουν η ευρωπαϊκή βιομηχανία ένα γήπεδο όπου παίζεται ένα παιχνίδι με καθαρούς κανόνες. Αλλά ακόμα και αν οι Ηνωμένε Πολιτείε, αν ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων δεχόταν αυτή τη συμφωνία, το Αμερικανικό Κογκρέσο θα απέριπτε μια τέτοια συμφωνία. Γιατί το Αμερικάνικο σύστημα ουσιαστικά λειτουργεί μόνο υπέρ των γηπέδων τα οποία δεν είναι ισόπεδα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε την ανεξαρτησία μας. Γιατί ποιος ξέρει τι θα φέρει το μέλλον, εάν αυτό το μέλλον βρίσκεται στα χέρια άλλων. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στην ε, πρωτοβουλία εκείνη την οποία ανέφερε ο πρόεδρος ε, και βεβαίως ε, θα μπορούσε κανείς να πει επιτέλους εάν όλη αυτή η εξέλιξη των μη πανδρομένων αεροσκαφών ήταν μια υπόθεση της προσωρινής αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και 15 χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες στην ίδια την Ευρώπη να καλύπτονται οι ανάγκες ε, από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελευταία δοκιμή. Όσον αφορά λοιπόν τους ε, λόγους που πως εδώ, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Αλλά είναι ένα διαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις ε, όσον αφορά τις ανάγκες μη επανδρομένων αεροσκαφών κυρίως καλύπτονται από αγορές στο εξωτερικό. Βεβαίως μπορεί κανείς να πει και Πού είναι το κακό. Ε, μη επανδρομένα είναι και δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβά. Κοιτάξτε όμως, εδώ υπάρχει το εξής. Πρώτον, εξαρτώματα πλέον από την ε, τεχνολογία του εκάστοτε προμηθευτή χώρας. Προμηθευτή, το θέμα δεν είναι και επανερχόμεθα εδώ στις ε, προηγούμενες παρατηρήσεις. Το θέμα δεν είναι να προσαρμοστούμε στους επερισμούς των ΗΠΑ όσον αφορά τη χρήση και την ε, περαιτέρω εξέλιξη. Αναφέρθηκε το παράδειγμα του Eurohawk ε, στη Γερμανία που δεν επιτρεπόταν η χορήγηση άδεια γιατί η ε, ευθύνη για την ενάρια αντίσταση αυτό ήταν απόλυτη αρμοδιότητα των ΗΠΑ και δεν μπορούσε να εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικότερα, στη Γερμανία. Και αυτό αφορούσε μέχρι και την απόδοση των υπολογιστών, τη διαδικτύωση και όλα τα σύναφη. Άρα δηλαδή αυτό είναι γεγονός και σημαίνει ότι όταν αγοράζει κανείς ε, εξοπλισμό στο εξωτερικό χάνει σε κάποιο βαθμό την ε, ανεξαρτησία του. Κατόπιν, το είπαμε, οι τεχνολογίες είναι επικαλυπτούμενες. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε μια τεχνολογία ε, μη επανδρομένων ή μαχητικών αεροσκαφών ε, πράγματι ή το ανώτατο επίπεδο επίπεδο αφορά ένα μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών στόχων. Το θέμα είναι ε, ότι κάποια στοιχεία υπάρχουν και στα μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια ολοκληρωμένη τεχνολογία και στρατηγική. Στην, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, πρέπει να σας πω ότι κατανείμαμε τα διάφορα συστήματα ανάλογα με τις ε, τεχνολογικές τους δυνατότητες, τις ε, βιομηχανικές ανάγκες και με τον τρόπο αυτό εντοπίσαμε τις επικαλύψεις. Προφανώς και υπάρχουν επικαλύψεις ε, όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και επικαλύψεις ανάμεσα στην αστική και την στρατιωτική χρήση. Αυτό που είπε δηλαδή ο κύριος Μάρσαλ. Κατόπιν τούτου υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά. Αυτό που παίζει ρόλο είναι, είναι η κάλυψη των αναγκών, υπάρχουν οι πρωτοβουλίες και οι δηλώσεις ε, των κατασκευαστών από πολύ σημαντικές ε, χώρες με αεροπορική βιομηχανία. Από την άλλη βέβαια πλευρά πρέπει να εναρμονιστούν οι ανάγκες έτσι ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική πρόοδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω και εγώ μέρα λόγια. Τα εξής. Έχουμε επιχειρηματολογήσει για τα βιομηχανικά, για τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά θα ήθελα να έχω τώρα μια πιο πραγματιστική προσέγγιση που είναι η πτυχή του προϋπολογισμού. Τη γνωρίζω πολύ καλά γιατί όταν ήμουν στην πολεμική αεροπορία είχα την ανάγκη να κάνω την δύσκολη αυτή διαμεσολάβηση ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες και τα διαθέσιμα κονδύλια. Ξέρω ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση, αλλά βλέπουμε ότι οι χώρες της Ευρώπης ε, μέσα σε αυτή την κρίση αναδιπλώνονται στον εαυτό τους αντί να προχωρούν σε καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους που είναι αυτό το οποίο εμείς υποστηρίζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. υπάρχουν λιγότερα χρήματα. Πρέπει να τα δαπανίσουμε καλύτερα και με πιο συντονισμένο τρόπο. Και εξάλλου, ανέφερα προηγουμένως τη μελέτη αυτή για το μέλλον στην Ευρώπη που λέει πράγματα πάρα πολύ συγκεκριμένα και απτά. Λέει ότι για μια περίοδο από το 2012 μέχρι το 2017 να εστιάσουμε στις ενέργειες τεχνολογικής έρευνας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δάπανο. Η έρευνα σε τεχνολογικό επίπεδο είναι κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια από το 2017 στο 2022 πρότεινα κάτι που είναι θεμελιώδης για μας να υπάρχουν προϊόντα επίδειξης ε, στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις επικοινωνίες των αεροσκαφών λοιπά, Και τα οποία μπορεί να κοστίσουν κάποιες εκατοντάδες εκατομμύριων ευρώ. Και μόνο από το 2022 όταν έχει υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ των χωρών στα προκατακτικά στάδια, τότε μπορούμε να έχουμε την εκκίνηση προγραμμάτων τα οποία θα δαπανίσουν δισεκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε φτάσει στο χρονικό σημείο που θα έχει περάσει ανάκαμψη η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και αναφέρω και μία, ε, μία περικοπή της πρότασης της Κομισιόν. Λέει ότι παρά τις περικοπές των κονδυλίων, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανούν περισσότερο συνολικά από ότι η Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία από κοινού. Όπως ξέρετε, η Ρωσία και η Κίνα αναπτύσσουν αεροπλάνα της πέμπτης γενιάς, αυτό δείχνει ότι και εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοια αεροσκάφη. Και θα ήθελα να έχω αυτή τη θετική νότα. Ευχαριστώ στρατηγέ μου. Ξεκινήσαμε κάπως αρνητικά και απεσιόδοξα, αλλά αυτό το οποίο είπατε είναι μια ελπιδοφόρα παρατήρηση και θα ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετέσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σωστά και πολύ καλά δώσει το περίγραμμα αυτών των θεμάτων και αυτά τα οποία λέμε για τα μαχητικά αεροσκάφη ισχύουν και για το σύνολο των αμυντικών θεμάτων, των ικανοτήτων μας και καταδεικνύουν τις βασικές έννοιες και κατευθυντήρες γραμμές που είναι οι σημαντικές για μας, δηλαδή το να προωθήσουμε μια στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, το να διατηρήσουμε μια βιομηχανική βάση και μια τεχνολογική βάση ευρωπαϊκή και επίσης ε, όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν σήμερα δείχνουν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αποφάσεις οι οποίες θα είναι εντυπωσιακέ στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά τουλάχιστον αυτό το Συμβούλιο μπορεί να είναι η απαρχή μιας διαδικασίας η οποία εν καιρό θα επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά στρατηγικών αποφάσεων, τότε νομίζω ότι θα είναι πολύ θετικό κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το προσδοκούμε. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια αν αυτό θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα ή όχι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και τις παρουσιάσεις σας. Θα είμαστε σε επαφή. Και ελπίζω να υπάρξει και επανάληψη αυτών των συζητήσεων μαζί σας. Bien, mesdames, messieurs, chers euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας με το επόμενο θέμα που είναι ένα εργαστήριο που αφορά την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε τη χαρά εδώ να έχουμε τέσσερις προσωπικότητες που θα μας ε, πλαισιώσουν με γνωστή ικανότητα για τα θέματα άμυνας. Το εργαστήριο αυτό εγγράφεται στα πλαίσια της έκθεσης της, Μαρία, της Μαριλένας Κοπά, της Επιτροπής μας, για την εφαρμογή της κοινής, εξωτε... της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Προφανώς εφέτος υπάρχει ιδιαίτερη σημασία για τα θέματα αυτά, γιατί εγγράφεται όλη αυτή η διαδικασία στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου που θα αντιμετωπίσει και θέματα άμυνας. Αλλά ακόμα και αν εμείς παραμένουμε πιστοί στην αρχική μας εντολή που είναι η εφαρμογή της ΚΕΠΑ, είναι φανερό ότι θα θέλαμε μέσω αυτής της ετήσιας έκθεσης να προχωρήσουμε και σε μια σειρά προτάσεων και να αντιμετωπίσουμε και θέματα για τα οποία είναι χρήσιμο να υπάρχει μια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Οι καλεσμένοι μας τους έχουμε γνωρίσει όλους σε διάφορες ευκαιρίες και έχουν εκφράσει την άποψή τους με δημοσιεύσεις ή με παρουσιάσεις σε σχέση με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να πριτανεύσουν στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για τις ε, πρόοδους που μπορούν να προκύψουν. Υπάρχουν πολλά λοιπόν άρθρα που έχουν δημοσιευτεί για τα θέματα αυτά, ιδίω η μελέτη του Ινστιτούτου Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως για τα θέματα των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το άρθρο αυτό είναι πολύ καλά συντεταγμένο. Έχουμε λοιπόν τέσσερις παρεμβαίνοντες, οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια και στο τέλος θα έχουμε την ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει. Έχω στα αριστερά το Τζο Κολμό, ο οποίος εκπροσωπεί το Ίδρυμα Έγμον, το Γιάννη Τέσσαου από το Ινστιτούτο Κάνεγκη στις Βρυξέλλες, τον Αντώνιο Μισιρόλη, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου για Αμυντικές Μελέτες στο Παρίσι και τον Αλεσάνδρο Μαρόνι από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στη Ρώμη. Είναι τέσσερις γνωστές λοιπόν και αναγνωρισμένες προσωπικότητες προτείνω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κόλμο. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και πρέπει να σας πω, ε, δεν θέλω να κρύψω ότι ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή για το μέλλον της ε, ΚΕΠΑ. Και πρέπει να σας πω ότι προσβλέπω στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου το Δεκέμβρη. Ελπίζω λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε σαφείς οδηγίες που θα μας δοθούν ε, για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Όχι μόνο όσον αφορά την ΚΕΠΑ, αλλά γενικά για την Ευρωπαϊκή Άμυνα υπάρχουν τρει τρεις τομείς, ε, τρία βασικά στοιχεία. Εγώ θα αναφερθώ στο πρώτο που έχει σχέση με τις επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο λοιπόν έχει ήδη καταθέσει κάποιες προτάσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς, μπορεί να, ε, πώς να πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ΚΕΠΑ και παράλληλα πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ταχύτατα και προληπτικά τις ε, σωστές ε, δυνατότητες. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ σε έξι υποσημεία. Το πρώτο αφορά τις επιχειρήσεις. Η επιχειρήση, δηλαδή το να αναπτύξει κανείς ε, μία επιχείρηση, αυτό είναι προνομία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, βεβαίως σε διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά νομίζω και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εάν ε, ανατρέξουμε στις επιχειρήσεις που έχουμε αναπτύξει μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγο να νιώθουμε απογοητευμένοι. Θα έλεγα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ε, σταδιοδρομίας μου είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μία ολόκληρη σειρά επιχειρήσεων είτε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, είτε του ΝΑΤΟ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε όλες τις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις που αναπτύξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φορά κατορθώσαμε να επιτύχουμε τους ε, στρατιωτικούς μας ε, στόχους. Και αυτό θα έλεγα είναι μοναδικό, μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα. Άρα δηλαδή έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε υπερήφανοι. Βεβαίως μετά, ε, μετά από την επιτυχία εύκολο είναι να πει κανείς ναι αλλά δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, ήταν επιχειρήσεις μικρής κλίμακας και ότι δεν είχαν και άμεση σχέση με την ασφάλεια. Δεν επαπειλεί η ασφάλεια. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού τα πράγματα δεν είναι έτσι και όχι μόνο από πολιτική σκοπιά. Σε πολιτικό λοιπόν επίπεδο ένα θέμα που πρέπει να τεθεί σχετικά με τις επιχειρήσεις είναι εάν πραγματικά επιτύχαμε ε, τους πολιτικούς μας στόχους και τους ε, στρατηγικούς μας και εδώ το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. διότι οι επιχειρήσεις αυτές ε, δεν ε, εμπνεύστηκαν τόσο πολύ από ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια. Με κάθε σεβασμό δηλαδή ε, σχεδιάστηκαν μέσα από μια διαφορετική νοοτροπία, την νοοτροπία του καλού. Δηλαδή ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάτι καλό, ας το κάνουμε. Κατόπιν τούτου Πράγματι, σημειώσαμε επιτυχία. Το πρώτο λοιπόν που μάθαμε είναι ότι αν θέλει κανείς να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ε, επιχειρήσεων ΚΕΠΑ, πρέπει κανείς να είναι σίγουρος ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης ε, ευρωπαϊκής στρατηγικής, ε, μια στρατηγική που καθορίσαμε το 2003. Δεύτερο θέμα, το να λειτουργεί κανείς προληπτικά οι επιχειρήσεις ε, στη Λιβύη και στο Μαλί απέδειξαν εκ νέου ότι οι προληπτικές ενέργειες πόσο μάλλον οι παρεμβάσεις, οι έγκαιρες παρεμβάσεις εντάσσονται στις διαρτρωτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τώρα πλέον οι επιχειρήσεις ad hoc έχουν ξεπεραστεί. Χρειαζόμαστε ε, μόνιμες ε, δομές, ε, τις μονάδες διοίκησης, αυτό είναι το πρώτο, και μετά ε, την ε, ανάπτυξη στρατευμάτων, μάχημων στρατευμάτων. Το 2003 νιώσαμε τέτοιο ενθουσιασμό όσον αφορούσε την επιχείρηση Άρτεμις στο Κονγκό και τα ταχύτατα αποτελέσματα που επιτύχαμε, έτσι ώστε αυτές τις δυνάμεις τις διαθέσαμε και μπορέσαμε να απελευθερώσουμε μία μάχη, μία ομάδα. Ενθουσιαστήκαμε τόσο πολύ που ε, αυτό μάλιστα συμπεριλήφθηκε ακόμα και στη συνθήκη. Και τώρα υπάρχει γενικότερα μία προσδοκία ότι όποια κρίση και αν ξεσπάσει η κρίση πρέπει να προσαρμόζεται στην ομάδα μάχης που είναι ε, η αντίστροφη εξέλιξη. Οι ομάδες ε, μάχης ε, είναι χρήσιμο εργαλείο στο βαθμό βέβαια που εντάσσονται στις ε, εφετρικές δυνάμεις. Εφεδρικές δυνάμεις χρειαζόμαστε ε, και για τα τρία όπλα, για τον εναέριο χώρο, χερσαίες δυνάμεις και θαλάσσιες δυνάμεις. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές του ΝΑΤΟ οι δυνάμεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι της ίδιας έκτασης όσο του ΝΑΤΟ, αλλά ούτε και μελιτές. Μπορούμε όλα αυτά να τα ε, καλύψουμε. Ναι, μπορούμε, το κάνουμε ήδη σήμερα μάλιστα. Και σε τελική ανάλυση αυτές οι εφεδρικές δυνάμεις πώς θα χρησιμοποιηθούν ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ε, αναπτυχθούν με βάση διαταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ. Εδώ μιλάμε γενικά για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε μια δεξαμενία αυτών των εφεδρικών δυνάμεων που ε, θα πρέπει να είναι οι πρώτες και που θα αναπτύσσονται για να διασφαλίζουν ότι θα καλύπτονται οι στόχοι τους οποίους ε, καλύπτουν, δηλαδή ε, οι στόχοι του Πίτερσμπουργκ. Το να υπάρξει λοιπόν μια τέτοια δεξαμενή εφεδρικών δυνάμεων, αυτό πλέον δεν ενδιαφέρει μόνο μία ή δύο χώρες. Ε, αφορά όλες τις χώρες και αυτό λοιπόν σημαίνει επίσης ότι αυτόματα υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη, επιμερισμός βάρους και κατά την άποψή μου πολύ σύντομα θα μιλάμε και για νέες οικονομικές ε, ρυθμίσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και η κριτική που ασκούμε κατά αυτό αυτής της ε, έννοιας των μάχημων δυνάμεων. Πάω τώρα στο τρίτο σημείο, στην ολιστική προσέγγιση. Αυτή η ολιστική προσέγγιση ε, έχει ε, περισσότερο σχέση με την διπλωματία, την άμυνα και την ε, ανάπτυξη. Εάν λοιπόν επιθυμούμε να υπάρχουν λύσεις διαρκείας, εάν επιθυμούμε να υπάρχει ένα πραγματικό πολιτικό αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε κατά νου και την οικονομική πτυχή του θέματος. Το λοιπόν που αναζητάμε τώρα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει κάποια μονάδα διοίκησης όπου όλες αυτές οι δυνατότητες θα συγκεντρώνονται που δεν είναι δηλαδή δεν πρέπει ε, να αντιγράψουμε αν θέλετε το shape του ΝΑΤΟ όχι κάτι άλλο εδώ αναζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο ε, θέλουμε να καλύψουμε και το οικονομικό στοιχείο και θέλουμε να το εντάξουμε στους υπάρχοντες θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Και φτάνω τώρα ε, στο τέταρτο στοιχείο ε, που ήθελα να αναφέρω. Ήδη αναφέρθηκα στο ΝΑΤΟ. Έχει φτάσει λοιπόν πλέον η στιγμή για να αντικατοστήσουμε τις ρυθμίσεις του Βερολίνου ε, στην ΚΕΠΑ και να βρούμε μία νέα έννοια Έχουμε τα τρία D του ΝΑΤΟ, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση, να μην υπάρχει επικάλυψη και ε, να υπάρχει αποσύνδεση από τα αγγλικά, από το D που υπάρχει στα αγγλικά. Εγώ τώρα όμως πάω σε μια καινούρια έννοια, όπου ε, πλέον το θέμα δεν είναι να έχουμε διασφαλισμένη πρόσβαση ε, στον ε, σχεδιασμό. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι πλέον τώρα να έχουμε τη μεταφορά των ε, υποδομών διοίκησης και ελέγχου και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ε, διαχείριση των κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΝΑΤΟ και από το ΝΑΤΟ ε, τα ΝΑΠΑΛΗ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με το ποιος αναλαμβάνει τη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό λοιπόν θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτο στοιχείο, ε, σχεδια... αμυντικός σχεδιασμός. Νομίζω όλοι οι εθνικοί αμυντικοί σχεδιασμοί τώρα σε όλες τις χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης κρίσεων. Το ένα είναι ότι οτιδήποτε και αν συμβεί Πολλοί ε, πίστευαν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα βοηθήσουν, αλλά αυτό πια πάβει να ισχύει ως αξίωμα. Τώρα στην Ουάσιγκτον έχουμε τον ε, πλέον ένθερμο υποστηρικτή της ΚΕΠΑ, αλλά αυτός ο υποστηρικτής περιμένει πλέον εμείς να αναλάβουμε τη, ταϊνία. να προβάλλουμε τις δικές μας δυνατότητες. Κατόπιν, σε όλες τις χώρες είχαμε εστιάσει την προσοχή μας σε τακτικές στρατιωτικές ικανότητες και είχαμε αγνοήσει τις στρατηγικές. Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί εμείς στην Ευρώπη για πάνω από 10 χρόνια ήμασταν σε θέση εκτός Ευρώπης να αναπτύξουμε για αρκετά χρόνια τόσες πολλές ένοπλες δυνάμεις. Άρα δηλαδή Έχουμε τις ικανότητες. Αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι οι στρατηγικές ικανότητες. Και οι επιχειρήσεις και στη Λιβύη και στο Μαλί κατέδειξαν με απόλυτη σαφήνεια ότι ο περιοριστικός παράγων για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η τεχνική, είναι ε, η στρατηγική. Έτσι λοιπόν στις χώρες μας αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι αλλάζει, μετατοπίζεται πλέον, ε, μετατοπίζονται οι προτεραιότητες του αμυντικού σχεδιασμού. Περνάμε σε στρατηγικές προτεραιότητες και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λυθεί σε εθνικό επίπεδο, άρα πρέπει να ε, συνενώσουμε τις δυνάμεις μας. Η λύση είναι να υπάρχουν υπάρχει κοινή αναζήτηση ε, λύσεων ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού. Και περνάω στο έκτο βασικό στοιχείο, τι προσβλέπω σε σχέση με το θερινό ε, Ευρωπαϊκό Σύμβουλο. Πολύ απλά να ε, προβληθεί έννοια ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι η άμυνα. Η άμυνα είναι καθοριστική για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, για το κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καθοριστική είναι η άμυνα όχι μόνο γιατί κοστίζει αλλά και γιατί αποτελεί επένδυση στην ασφαλειά μας. Και νιώθω την εξής ελπίδα ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα ε, λάβει ε, μια καλύτερη προσέγγιση κατευθύνσεις από πάνω προς τα κάτω και πρέπει να σας πω ότι είμαι ευγνώμων σε αυτό το κοινοβούλιο γιατί εσείς αυτό ανέκαθεν κάνετε. Δηλαδή ανέκαθεν αποδίδετε σημασία στην άμυνα και τη λαμβάνατε σοβαρά υπόψη σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τεσσό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα να πάρω το λόγο ενώπιον αυτό της Επιτροπής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν ε, αναφερόμαστε στην ΚΕΠΕ, Έχω την εντύπωση ότι μας λείπει ένα σημείο αναφοράς για να αποφασίσουμε αν είναι καλή ή κακή. Όταν βλέπουμε την ΚΕΦ στα πλαίσια των πολιτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη για να μπορέσει να μιλήσει με μία φωνή, η ΚΕΠ διαπιστώνουμε ότι είναι καλύτερη από ό,τι φημολογείται ότι είναι ε, πηγαίνει σε αποστολές και αποτελεί προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Όταν όμως εξετάζεται την ΚΕΠΕ ως έχει, ε, οι στατικές ανάγκες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και θα αντιμετωπίσει και στο μέλλον θα διαπιστώσουμε ότι είναι ανεπαρκή σε μεγάλο βαθμό και το θέμα είναι ε, πώς συγκεράζουμε τα δύο αυτά σημεία αναφοράς και πώς θα μπορούσαν να έχουν και κάποιο νόημα εν ώψη της επερχόμενης διάσκεψης κορυφής. Βασικά θα με απασχολήσουν οι στατικές ανάγκες και οι πλημελείς ε, επιδόσεις της ΚΕΠΕ. Ποιες είναι οι στατικές ανάγκες. Στην πραγματικότητα η ΚΕΠΕ κατά βάση αφορά το ερώτημα τι κάνουν οι Ευρωπαίοι και δεν κάνουν οι Αμερικάνοι. Σε μεγάλο βαθμό βασιζόμαστε στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας για να προστατεύσουμε όχι τη φυσική μας ασφάλεια, Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι πλέον βασικό θέμα, ότι η Ανατολική Ευρώπη το βλέπει διαφορετικά. Το θέμα αφορά την προστασία των παγκοσμίων ε, συμφερόντων ασφαλείας. Εμείς παίρνουμε μέρος σε ένα μικρό βαθμό, αλλά σε μεγάλο βαθμό παρέχεται από κάποιον άλλον. Εμείς βασιζόμαστε σε μια φιλελεύθερη ε, τάξη, σε μια πρόσβαση σε αγορές, σε γραμμές επικοινωνίας και παίζουν ηγετικό ρόλο σε επίπεδο σειράξεων σε όλο τον κόσμο, γιατί επηρεάζουν όλη την οικονομία. Βασιζόμαστε λοιπόν στις ΗΠΑ για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση αυτή για δύο λόγους, γιατί οι επιχειρήσεις αυτές ευθύνουν όλο και περισσότερο. Ξέρετε ότι οι ΗΠΑ περιορίζουν περιορίζουν την επιρροή τους σε πολλά ε, μέτωπα και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες, αλλά δεν είναι βιώσιμο γιατί μειώνει τις πολιτικές μας δυνατότητες να επηρεάσουμε τα πράγματα. Αυτό έχει σχέση με τις φυσικές μας ανάγκες, αλλά και με το θέμα της ε, πολιτικής μας ισχύω και δυνατότητας επιρροής. Πόσο θέλουμε, πόσο χρειαζόμαστε. Υπάρχουν έξι σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Τι περιμένουμε δηλαδή από την επερχόμενη διάσκεψη κορυφής. Το πρώτο αφορά την αλλαγή νοοτροπίας. Η αλλαγή νοοτροπίας θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε το στρατηγικό δίλημα ενώπιον του οποίου βρίσκεται η Ευρώπη. Ότι βρίσκεται σε ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να στηρίξει και δεν μπορεί να εγγυηθεί, ότι χρειάζεται άλλους. Πολύ συχνά απευθύνομαι σε διαφορετικά ακροατήρια στην Ευρώπη και λέω και συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει απόλυτη συνείδηση αυτού του γεγονότος. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα, δηλαδή να Υπάρχει η απαιτούμενη οτροπία για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Όχι στα πλαίσια της ρητογική μιας διάσκεψης κορυφής, αλλά στα πλαίσια της συνειδητοποίησης μιας ανάγκης. Το δεύτερο, η ε, δεύτερη ελπίδα μου έχει σχέση με την κοινή μας άποψη. Όλοι διαμαρτυρόμαστε για την απουσία πολιτικής βούλησης Υπάρχουν ορισμένοι στρατηγικοί στόχοι, αλλά πολύ σπάνια βρίσκεται ο κατάλληλος τρόπος ε, για να εφαρμοστούν. Όλα αυτά είναι προβλήματα, αλλά το υποκείμενο θέμα για μένα και το βασικό αίτιο είναι ότι δεν υπάρχει μία κοινή προοπτική, ένας κοινός τρόπος αξιολόγησης της κατάστασης. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς πληροφόρησης, ε, ε, αξιολόγησης και να δημιουργήσουμε το ίδιο αυτό της κοινή άποψης, ε, αλλά στην πραγματικότητα δεν κατανοούμε τι θα είναι επικίνδυνο, τι θα μπορούσε να διακυβεύσει την ασφάλειά μας. Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές εμπειρίες που έχουμε αναπτύξει το παρελθόν και τι πολιτικέ διαφορέ μεταξύ των χωρών μελών. Εάν θέλετε, θέλουμε όμω να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να καταβάλουμε μία επιπλέον προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η κοινή αντίληψη. Αυτό που ελπίζω λοιπόν είναι αυτή η κοινή μηχανισμοί, ε, αυτά τα μέσα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθεί, ε, για να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς είναι κάτι που πραγματικά θα επιθυμούσα να γίνεται. Και αυτό με οδηγεί στο τρίτο σημείο της παρέμβασής μου. Βέβαια, δεν ε, ε, ηχεί καλά το να λέγεται κάτι τέτοιο στις Βρυξέλλες, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται περισσότερες συναντήσεις. Ε, οι Υπουργοί Άμυνα είναι τα παραπέδια της ΚΕΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν τα πράγματα να αλλάξουν, θα πρέπει τα πράγματα να τίθενται πιο συχνά επιτάπητος. Αυτό είχε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που νομίζω ότι θα πρέπει να συναντάτε τουλάχιστον ε, μία φορά, να μην είναι αμυγός ένα Υπουργείο Άμυνας, αλλά ε, να συναντώνται και να συζητούν θέματα που είναι στην ημερησία διάταξη ε, και ένα από τα θέματα θα είναι και η αξιολόγηση των όσων έχουν γίνει. Όπως είπε ο, ε, ο πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα σε όσο γίνεται πιο υψηλό επίπεδο. Το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι κάτι που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από μερικούς μήνες όταν πρότεινε ένα έγγραφο για το θέμα του κοινού τρόπου αντίληψης ε, των διαφόρων θεμάτων στην Ευρώπη, ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μία πιο συνδυασμένη στρατηγική αντίληψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων είπε ότι η Υπουργή Οικονομικών θα μπορούσαν να συμφωνήσουν για ένα δημοσιονομικό εξάμεινο <clears throat> που θα συγκρίνουν στοιχεία που αφορούν ε, τις δαπάνες. Ε, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια πιο κοινή αντίληψη αλλά και μια γενικότερη ιδέα για το τι κάνουν οι άλλοι. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να υποβάλουν τα προγράμματά τους αιτιολογώντας γιατί τα κάνουν σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να μιλάνε για αυτά και να δημιουργούν μια δυναμική για να καταλήγουν οι δυνατόν σε μερικά συμπεράσματα. Το πέμπτο σημείο έχει σχέση με το ιστορικό κανονισμό. Νομίζω ότι όλοι μας ή σχεδόν όλοι μας πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις του μέλλοντος και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό οι συμμαχίες των αυτών που θέλουν να συμμετάσχουν. Δεν είναι λοιπόν όλες οι χώρες οι οποίες θα συμμετέχουν πάντα σε όλες τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, μόνο κάποιες χώρες, θα, κάποιες ομάδες θα είναι διαθέσιμες για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα όμως. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι στους εσωτερικούς κανόνες λήψης απόφασης, ώστε όλοι μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις που θα γίνουν από μερικές μοναχά χώρες. Αυτό δόθηκε, ένα καλό παράδειγμα δόθηκε στο, στη Λιβύη. Οι περισσότερες χώρες δεν θέλαν να συμμετάσχουν, αλλά όλες υποστήριξαν την διαδικασία αυτή, είπαν ναι στο ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ευελιξία για κάποιες χώρες να μην συμμετέχουν, αλλά να μην εμποδίσουν τη δράση των υπολείπων. Η δεύτερη συνέπεια είναι, να δω τα χαρτιά μου μια στιγμή, είναι ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η διαδικασία λήψης απόφασης. Φυσικά όταν ζητάμε από τα κράτη-μέλη, από τα 28 κράτη-μέλη να συμβάλλουν σε κοινά στοιχεία τα οποία συμμετέχουν στην ε, επιχειρησιακή ικανότητα, αλλά μόνο μερικά κράτη χρησιμοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία, τότε αν αυτό γίνεται συνέχεια, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία ορισμένων χωρών. Πρέπει να υπάρχει κάποιο σύστημα αντιστάθμισης, ώστε όλες οι χώρες έχουν το ενδιαφέρον να διατηρήσουν το, τη χρηματοδότηση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι μόνο μερικές χώρες χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστή σκέψη για τα θέματα αυτά. Και το τελευταίο μου ε, σχόλιο, και εδώ πολλές φορές ε, αντιμετωπίζω γέλοτες από το ακροατήριο, ακούσαμε ότι δεν είναι πιθανή η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη και παρόλα αυτά παρά τις δαπάνες που γίνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, δεν έχουμε την απαραίτητη στρατηγική ικανότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι η λύση σε αυτό είναι μεγαλύτερη αποδοτικότητα, μεγαλύτερη συμμετοχή όλων και πιο αποτελεσματικός, αποτελεσματική χρήση. Τα χρήματα που μπορείτε να εξοικονομήσετε από την θέση ε, σε, από την κοινή χρησιμοποίηση όλων αυτών των ε, αμυντικών στοιχείων είναι πολύ μεγάλη και αυτό μας δίνει την απαραίτητη ικανότητα που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό, αυτή την ε, συνένωση των προσπαθειών μας και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να χρειαστεί να δαπανίσουμε και περισσότερα σε ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στον εαυτό μας αν η ανάγκη να έχουμε περισσότερες υπηρεσίες ασφάλειας σε μια ασταθή παγκόσμια κατάσταση είναι απαραίτητη και αν γίνεται πιο δύσκολος ο κόσμος, γίνεται πιο πολυπολικός και πιο ασταθής. Αν λοιπόν είναι πιο δύσκολη η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, τότε θα πρέπει να δαπανούμε λίγο περισσότερο στην άμυνά μας και ελπίζουμε πιο ευφύη τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέγει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό πιστεύω. Ο κύριος Μισηρόλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Εγώ θα έχω μια κάπως εμπορικού χαρακτήρα παρέμβαση. Έχουμε παρουσιάσει το Ινστιτούτο με μια έκθεση στην Στρατιωτική και Πολιτική Επιτροπή σε σχέση με τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για το μέλλον αυτών των ενεργειών. Έχω φέρει κάποια αντίγραφα αυτή τη έκθεση που μπορείτε να δείτε εδώ. Μπορείτε φυσικά να απευθυνθείτε σε εμά γραπτό αν θέλετε να έχετε περαιτέρω αντίγραφα. Εγώ θα συνοψίσω μόνο τα κύρια σημεία τη έκθεση. και θα είμαι λίγο σύντομος και λίγο επιφανειακός στην παρουσίαση αυτή. Θέλαμε να εστιάσουμε στο μέλλον περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και ίσως δεν πρέπει να εστιάζουμε υπερβολικά στο τωρινό χρονικό σημείο. Μας, ε, το σημείο αναφοράς μας είναι το 2025 γιατί αυτό είναι ένα χρονικό ορόσημο σε σχέση με τις ικανότητες Ευρώπης στο στρατιωτικό επίπεδο. Όλα αυτά βέβαια είχαν θεσπιστεί πριν από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ενδεχομένω θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και τα στοιχεία αυτής της δημοσίευσης μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν, βλέπω δεν ξέρω αν βλέπετε τα, τις διαφάνειες. Η βασική ιδέα ήταν να ξεκινήσουμε με μια θετική αναγνώριση όλων αυτών που έχουμε επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέποντας συγχρόνως και τους περιορισμούς και τις ελλείψεις της προσέγγισή μας για την ανάπτυξη στρατιωτικής ικανότητας. Και εδώ περιλαμβάνεται το γεγονός ότι είναι ακόμα κατακαιρματισμένο το τοπίο σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει. Αυτά είναι τα κύρια επιτεύγματα των προηγουμένων ετών. Δεν πρόκειται να σταθώ σε αυτό. Και εδώ είναι οι κύριες ελλείψεις που έχουμε εντοπίσει στην εκθεσή μας. Και εδώ υπάρχει μια υφέρπουσα αποστρατικοποίηση. Θυμάστε αυτά που είχε πει ο Bill Gates πριν από δύο χρόνια. Και το γεγονός ότι αυτό σημαίνει και μείωση της βιομηχανικής ικανότητας στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Μια δυναμική αστάθεια και συστημική αλληλεξάρτηση στο παγκόσμιο σύστημα, την ανάδυση νέων περιφερειακών δυνάμεων, ιδίως στην Ασία, τον κεντρικό ρόλο των ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση που κάνει την ε, ε, η γειτονιά μας θα είναι πιο κοντά σε εμά από το Μάλι στην Σομαλία, στο Αφγανιστάν και επίσης εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναδιατυπώσει τα στρατηγικά της συμφέροντα, κάτι το οποίο αναφέρει και το άρθρο 26 της Συνθήκης Λισαβόνας, που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να λέει περισσότερες λεπτομέρειες και φαντάζομαι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πρέπει να είναι και η απαρχή αυτών των συζητήσεων. Έχουμε εντοπίσει μερικές τέτοιες ε, περιπτώσεις που πρέπει να σκεφτούμε και φυσικά και εσείς θα μπορέσετε να δώσετε τα δικά σας φώτα για τα θέματα αυτά. Τα ανοιχτά ερωτήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το Δεκέμβριο είναι τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε μια σειρά από δρόμους που θα οδηγήσουν σε καλύτερη ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων. Δεν είναι αλλοαποκλειόμενοι αυτοί οι δρόμοι, έχουν σωρευτικό χαρακτήρα οι πρόοδοι σε αυτές τις επιλογές. Είναι όλα αυτά ε, επιλογές που δεν είναι αποκλείουσε στις άλλες επιλογές. Μιλήσαμε για εδραίωση, για βελτιστοποίηση, για καινοτομία περιφερικοποίηση και ολοκλήρωση. Καταρχήν, η ενοποίηση, η παγιοποίηση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη στρατιωτική ικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τα απεπαλαιωμένα στοιχεία που έχουμε στην Ευρώπη για να κάνουμε εξοικονόμηση και μια τέτοια δυνατότητα για να απαλύνουμε και τον κοινωνικό αντίκτυπο θα είναι πάντα να χρησιμοποιήσουμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης και τα διαφορετικά ταμεία τα οποία βρισκόνται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα κάνει κάποιες αναφορές σε αυτή τη δυνατότητα. Προτείνουμε επίσης να υπάρξει μια κάποια στρατιωτική επισκόψη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια είναι ακόμα μια προκατακτική άσκηση, κάτι ανάμεσα σε μια πράσινη βίβλο και σε μια άσπρη βίβλο. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εργαστεί ιδιαίτερα για μια λευκή βίβλο. Κάποια κράτη-μέλη βέβαια θα έχουν αντίρρηση σε μια λευκή βίβλο γιατί πολλές φορές έχει ένα ιδιαίτερα περιοριστικό χαρακτήρα σε σχέση με τις ε, επιλογές ενώ μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε τη γενική μορφή της αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά μπορεί να είναι μια χρήσιμη άσκηση γιατί θα δώσει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αυτή την άσκηση και να καταγράψουν τις ικανότητες που υπάρχουν και τις ανάγκες του μέλλοντος. Ο δεύτερος δρόμος είναι βελτιστοποίηση, βελτιστοποίηση για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο αντιοτικό τομέα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα, οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη μελλοντικών δυνατοτήτων. Και επίσης για να μεταλαμπαδεύονται οι καλύτερες πρακτικές, οι νέες ε, αντιμετωπίσεις για την προμήθεια οπλικών συστημάτων που μπορούν να εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτος δρόμος είναι η καινοτομία, η ενίσχυση της στρατιωτικής τεχνολογίας και να ξεπεράσουμε το κίνδυνο της αποβιομηχανοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί η καινοτομία οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και σε τεχνολογική πρόοδο. Η χρηματοδότηση έρευνα και τη ανάπτυξης είναι απαραίτητη και οι εξοικονομίες οι οποίες γίνονται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να μεταφερθούν σε κοινέ ευρωπαϊκές επενδύσεις. αυτό είναι ένας πολύ χρήσιμος δρόμος για να προχωρήσουμε. Και μπορούμε να έχουμε στοχευμένες λύσεις για να μπορέσουμε να δανειστούμε ιδέες από προηγούμενες ενέργειες όπως παραδείγματος αυτά που γίνονται στο ΝΑΤΟ για τα AWACS ή από άλλους χώρους πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα λεγόμενα ε, ομόλογα έργων. Τέταρτον, η καλύτερη περιφερικοποίηση για να έχουμε μεγαλύτερο εύρος και μεγαλύτερο βάθος της επιχειρήσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συμπλέγματα χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεργάζονται ήδη διμερώς μεταξύ τους ή μινιπολικά όπως λέγεται σε ακαδημαϊκούς κύκλους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εξοικονόμηση Αυτές οι μορφές συνεργασίας όμως μπορούν να τεθούν σε κοινό πλαίσιο ώστε αυτές οι νησίδες ε, μπορούν να γίνουν ένα νησιωτικό σύμπλεγμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων. Τέταρτο, πέμπτο αλλά όχι τελευταίο είναι οι κινήσεις προς περισσότερη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση που θα αυξήσουν το βάθος της ικανότητάς μας και την βιωσιμότητά του. Υπάρχουν πολλές ιδέες οι οποίες έχουν διατυπωθεί στο άρθρο μας για τα διδάγματα που μπορούμε να ε, λάβουμε α, για τις ε, αεροπορικές επιχειρήσεις της Ευρώπης να υπάρχει κάποιος στόλος ο οποίος θα μπορεί να καλύπτει τις ενέργειες οι οποίες αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραγωγή χάρη έξω από τις ακτές της Σομαλίας. Όλα αυτά αποτελούν το να, τονίζουν την ανάγκη να έχουμε ένα νέο αριθμό κυρίων στόχων για το 2025 και να έχουμε καλύτερο συγχρονισμό των εθνικών κύκλων προμήθειας και ανάπτυξη των οπλικών συστημάτων μεταξύ τους για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εν κατακλείδη, οι Ευρωπαίοι χάνουν την κυριαρχικότητά τους εάν δεν ενοποιήσουν, δεν βελτιστοποιήσουν, δεν καινοτομήσουν και δεν προχωρήσουν σε περιφερικοποίηση και ολοκλήρωση των στρατιωτικών της ικανοτήτων οι πολιτικές πρόκλησεις, που έχουμε απαιτούν μια συνεχή και συστηματική επανεξέταση των ε, δυνατοτήτων μας. Ένα από τα κύρια αποτελέσματα η, της έκθεσής είναι ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε με σε απομόνωση τις στρατιωτικές προκλήσεις. Όλο και περισσότερο θα πρέπει να λειτουργούμε σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών εργαλείων πέραν και των στρατιωτικών εργαλείων όλες οι πτυχές Φυσικά έχουν και μια στρατιωτική διάσταση σε ό,τι αφορά την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συνεργασία. Και πάλι τα διδάγματα μπορούν να μεταλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα πολιτικής και σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο όλοι αυτοί οι δρόμοι πρέπει να συνενωθούν μεταξύ τους και να αντιμετωπιστούν σωρευτικά, αλλά χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις για να γίνουν πραγματικότητα οι δηλώσεις, οι οποίες ακούγονται πολλές φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά το τελικό μας σημείο και συμμερίζονται πολύ πιστεύω αυτή την απόψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης και όχι το σημείο άφηξης για να μπορέσει να ξεκινήσει ένας κύκλος πολιτικών ενεργειών και συντονισμού που να μπορέσει μέσα στα όρια τα οποία υπάρχουν να είναι το αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όχι για την άμυνα μονάχα, αλλά γενικά για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Well, first of all, uh, let me thank the European... Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης. Οι παρατηρήσεις μου που θα συμπληρώσουν αυτές των προηγούμενων μιλητών αφορούν ε, θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην ε, στρατιωτική βιομηχανία και το τι αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το πρώτο σημείο αφορά μια διευκρίνηση για το γεγονός ότι είναι καλύτερα να μιλάμε για μια όχι για βιομηχανία όπλων, αλλά για βιομηχανία άμυνας, γιατί σήμερα η βιομηχανία παράγει ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, σε επίπεδο τεχνολογίας, σε επίπεδο αύξησης ικανοτήτων κτλ. Το δεύτερο, αποτελείται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων εταιριών και με ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι δηλαδή σαν ένα τραπέζιο. Η βάση λοιπόν αφαίρεται στο γεγονός ότι αυτό υφίσταται στις ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει ε, παροχή και σε υπηρεσίες ασφαλείας και στις στρατιωτικές δυνάμεις αλλά και σε ε, ε, πολίτες. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσοι έχουν ή μη μικρές προσαρμογές ανάλογα με τη χρήση που θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή ο ευρωπαϊκό Οργανισμός Άμυνας αναφέρεται σε μια ευρωπαϊκή τεχνολογική βάση και αμυντική βάση. Δεύτερο θέμα, το δεύτερο αφορά τη συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πήγε ξεκίνησε σε εθνικό επίπεδο και παρέμεινε έτσι για πολλές δεκαετίες. Πολλές χώρες μέλη συνεπώς συνεχίζουν να πιστεύουν, να τη θεωρούν ότι είναι κάτι εθνικό στην πραγματικότητα, όμως είναι παγκόσμιο για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η αυξημένη ε, εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές αγορές. Ξέρετε ότι οι δαπάνες σε επίπεδο ευρωπαϊκό μειώνονται, αλλά οι αμυντικές δαπάνες εκτός Ευρώπης αυξάνονται. Συνεπώς η εθνική αμυντική πολιτική θα πρέπει για να επιβιώσει να χρησιμοποιήσει άλλες αγορές. Ινδία, Βραζιλία, Κατάρ, Σαουδική, Σαουδική Αραβία, Ιωνισία, ε, Κατάρ. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση επειδή πολλές από αυτές τις χώρες θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους βιομηχανική ε, αμυντική βάση, ζητώντας από τις ευρωπαϊκές εταιρείες ε, να παράγουν τοπικά ή να μεταφερθεί, ζητά να μεταφερθεί τεχνολογία από την Ευρώπη σε αυτές τις χώρες. Μολονότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προσεκτικά από την πτυχή της βιομηχανία και της ασφαλείας, θα πρέπει ε, να δώσουμε τη δυνατότητα συνεχικούς προμήθειας των ενόπλων δυνάμεων. Πάρα πολλές φορές το ίδιο προϊόν εξάγεται σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Το δεύτερος λόγος που οι πολιτικές αυτές είναι περισσότερο παγκόσμιες είναι επειδή έχει ένα παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα η αλυσίδα της ε, τροφοδοσίας. Πολλοί επενεργούν ως ε, ανάδοχοι, ως υπεργολάβοι συμβάλλοντας στο ευρύτερο σύστημα. Σήμερα η αλυσίδα αυτή αποκτά ένα, όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα. Και οι προμηθευτές είναι οι περισσότεροι μη Ευρωπαίοι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο ανταγωνιστικές λόγω χαμηλότερου κόστους ή γιατί οι τοπικές κυβερνήσεις ε, παραχωρούν ένα μέρος ε, της παραγωγής στα πλαίσια ενός τοπικού προγράμματος. Μερικά, μερικά ε, εξαρτήματα ή ε, πρώτες ύλες παρέχονται από μη ευρωπαϊκή εταιρείες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου από άποψη ασφάλειας και άμυνας. Η πλατφόρμα που απαιτείται από τις ευρωπαϊκές ενόπλες δυνάμεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ευρωπαϊκή γιατί παρέχεται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να εξαρτάται από εξαρτήματα, πρωτεσίλες και τεχνολογίες από μη που προέρχονται από μη ευρωπαϊκές πηγές. Με λίγα λόγια, ο Ευρωπαίος προμηθευτής μπορεί να διαπιστώσει έλλειψη ε, ε, εξαρτημάτων ή οτιδήποτε. Το τρίτο θέμα αφορά την αυξανόμενη σημασία των τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές, οι διτές αυτές τεχνολογίες συνδέουν το στρατιωτικό με το πολιτικό σκέλος σε όλο τον κόσμο για παράδειγμα, οι πωλήσει μπορούν να γίνουν είτε στην Frontex, είτε στην ε, αεροναυτική βιομηχανία στι ΗΠΑ κτλ. Πρόσφατα διαπιστώθηκε μια συγκεκριμένη εξέλιξη. τεχνολογική εξέλιξη έχει, ε, δείχνει σημεία ιδιαίτερης επιτάχυνσης. Συνεπώς, η τεχνολογική ανωδική τάψη στάση η σχέση μεταξύ του πολιτικού και στρατιωτικού τομέα έχει αυξηθεί. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτώμεθα περισσότερο από τους πολιτικούς προμηθευτές, μη στρατιωτικού προμηθευτές, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, την εξάρτηση από τους ε, νέες αγορές, η σημασία διετής τεχνολογίας και η εξάρτηση αυτό σε συνδυασμό με ε, την εξάρτη, με, ε, ε, σε συνδυασμό με το θέμα των προμηθειών έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. To the European integration of uh, DTB. <coughs> vis a -vis the globalization της παγκοσμιοποίησης ο εξευρωπαϊσμός της πολιτικής είναι μια καλύτερη επιλογή γιατί εξασφαλίζει μια καλύτερη ασφάλεια προμηθειών γιατί οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες είναι περισσότερο αλληλεξαρτώμενες σε σχέση με άλλες μη ευρωπαϊκές εταιρείες αφού αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών ε, εταιριών μέσω, οικονομία, μέσω οικονομίας ε, κλίμακας και συμμετέχει στην όλη την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκληρωση. Αυτό είναι εφικτό λόγω, ε, εξαιτίας πέντε βασικών λόγων. Πρώτον, οι δαπάνες παραμένουν σημαντικές σε αυτό το τομέα η Ευρωπαϊκή Πολιτική περιλαμβάνει πολύ ανταγωνιστικές εταιρείε καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι 40 από τις βασικότερες εταιρείε στον τομέα αυτό είναι ευρωπαϊκές. Τρίτον, ο τομέα αυτό έχει ένα κύκλο εργασιών, εργασιών που ανέχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ με 47.000 απασχολούμενος. Υπάρχει άλλος λόγος ότι υπάρχει ένα δίκτυο ε, συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας. Υπάρχουν προγράμματα όπως το Eurofighter ή το πρόγραμμα για τα ελικόπτερα. Τέταρτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε δύο σημαντικές οδηγίες που αφορούν το αμυντικό πακέτο. Μόλις εφαρμοστούν θα δημιουργήσουν ένα ε, νομικό πλαίσιο. Τέλος, υπάρχουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν σημαντική αγορά σε διάφορες αγορές και από την άποψη του μεσγκριδίου και από την άποψη των ε, ικανοποίητων. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα διακρατικών ε, εταιριών όπως η βιομεκάνικα που θα μπορούσαμε να την παραθέσουμε ως παράδειγμα. Το τελευταίο μου σημείο αφορά τις προκλήσεις στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της πολιτικής. Μία πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική είναι κάτι δύσκολο και δεν υπάρχουν βεβαιότητες ότι θα επιτύχει. Η Στις περισσότερες ε, περιπτώσεις ε, ακολουθείται η αμυντική πολιτική μέσα σε εθνικά πλαίσια, παρόλο που δίνονται όλο και λιγότερα κονδύλια για τις Είναι θέμα ασφάλειας προμηθειών, αλλά και θέμα του να διατηρηθούν σε μια χώρα εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι κάτι που καθίσταται σαφές από την ε, έλλειψη προθυμίας από πλευράς πολλών κυβερνήσεων να κάνουν κάτι μόνο ότι έχουν αλλάξει πολλές, ένα μεγάλο μέρος της εθνικής νομοθεσίας. Από την άλλη πλευρά δεν είναι πεπισμένοι όλοι για τον στόχο του να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αγορά, αμυντική αγορά. Αυτό καθίσταται σαφές από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το υπάρχουν, ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 και τα περισσότερα αρχίζουν και φθήνουν. Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί προετοιμάζουν το έδαφος για μελλοντικά κοινά προγράμματα προμηθειών. Το 87% των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης έλαβαν χώρες εθνικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν αποτελεί συνταγή για να συνεχιστεί αυτός ο κατακαιρματισμός που παρατηρείται και κατά συνέπεια για, τον, ε, για τη συνέχεια της αναποτελεσματικότητας της βιομηχανίας αυτής. Το συμπέρασμά μου είναι ότι να γνωρίζουμε ότι οι τρεις αυτοί τομείς της ε, Ευρωπαϊκής Βάσης Άμυνας θα συμπεριληφθούν στο, στη διάσκεψη κορυφής ε, του Δεκεμβρίου, γιατί τα πράγματα, οι τομείς αυτοί δεν επηρεάζουν ο ένας τον άλλον με άμεσο τρόπο. Η ειδική πολιτική έχει, ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί επηρεάζει την προσέγγιση προ οποιαδήποτε διαδικασία τη Ευρώπη στον τομέα τη άμυνα, λαμβάνοντα υπόψη την ε, παγκοσμιοποίηση της πολιτικής αυτής θα έλεγα ότι είναι προς το συμφέρον οποιασδήποτε εθνικής πολιτικής να επιτύχει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε αυτό το τομέα και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο θα δώσει μία πολιτική εντολή να συνεχιστεί αυτή, να δοθεί συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία. Η πλήρης εφαρμογή των οδηγιών είναι αναγκαία μέσω του, της αύξησης, ενδυνάμωσης, του ελέγχου ε, των κυβερνήσεων αυτών που ε, δεν, δεν παρουσιάζουν, ε, δεν έχουν προθυμία να συμμορφωθούν και ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός οδηγικός χάρτης θα είναι αναγκαίος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το κατακαιρματισμό των δραστηριοτήτων έρευνα και τεχνολογία. Συμπεριλαμβαντικά υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσεις στη διαδικασία αυτής της παγκοσμιοποίηση πολιτικής. Κάτι δύσκολο αλλά εφικτό και πρωτίστω αναγκαίο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour... Euh, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τα πλήρη σχόλια που μας δώσατε σε σχέση με τα τρία βασικά καλάθια κατά κάποιο τρόπο, επιχειρήσεις, ικανότητες και βιομηχανία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Μαριλένα Κοπά που είναι η συγητρία μας για την ετήσια έκθεση, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε ο κ. Τεσό, ιδίω για την έκθεση αυτή. για τα Υπουργεία Άμυνας που είναι τα ορφανά της ΚΕΠΑ Εγώ θέλω να σας αναφέρω μια ιστοριούλα που αναγκάζομαι να την ε, υπενθυμίσω. Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στο Δουβλίνο το Φεβρουάριο του 2013 που ήταν μόνο οκτώ χώρες οι οποίες είχαν εκπροσωπηθεί και όπου είχαν πάει πολλοί στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ που ασχολιόταν με θέματα ίσονα συνεργασία με την Ουκρανία κτλ. Εκεί ήταν όλοι οι υπουργοί λοιπόν των ευρωπαϊκών κρατών Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ πελόδοξοι, αλλά και ρεαλιστές για τα θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας υπάρχουν, υπάρχει πολλής δρόμος ο οποίος πρέπει να γίνει και από τους ε, υπουργούς των κρατών μελών Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα δώσω την προεδρία στον κύριο Σοφοκλέους και θα ζητώ συγγνώμη, αλλά σας ευχαριστώ για την συμβολή σας στη συζήτηση και κατά 90% εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που έχετε πει και θα δώσω το λόγο στη Μαριλένα Κοπά. Euh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και τους ε, συμμετέχοντες στο πάνελ για τις παρεμβάσεις τους που είναι πολύ σημαντικές. Η ετήσια έκθεση είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε με πιο συνολικό τρόπο τα θέματα άμυνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτά για ένα εξάμεινο που σίγουρα τα θέματα άμυνα θα είναι στη μέση διατάξη του Συμβουλίου. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα στο Συμβούλιο για, σε ό,τι αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου. Η δική μου πρόθεση είναι να ακολουθήσω την ε, δομή του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι οι ικανότητες, οι προοπτικές και η βιομηχανία. Για πολλούς φαίνεται πολυτέλεια η συζήτηση της άμυνας και της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για μένα όμως αυτό μου φαίνεται λαθασμένο και συμμερίζουμε αυτά που λέτε ότι είναι σημαντική η άμυνα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και μια καλύτερη επικοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ανταλλάσσουμε απόψεις μεταξύ μας, αλλά εμείς είμαστε ήδη πεπισμένοι για τα θέματα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη εκστρατεία επικοινωνίας από τη δική μας πλευρά, αλλά ελπίζω και από την Κομισιόν, από τα αμυντικά Ινστιτούτα, και εδώ σκέφτομαι για το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, όλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε ότι χρειάζεται καλύτερο σχεδιασμό τη συζήτηση για μια εν καιρό μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής άμυνας στα επόμενα 2-3 χρόνια. Πρέπει τα θέματα αυτά να είναι στη μεσή διαταξή. Δεν μπορεί να είναι μια συζήτηση ad hoc. Δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο επανέρχεται σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η άμυνα είναι κάτι που δεν έχει πρώτη στη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το λαθασμένο μήνυμα που δίνουμε. Τρίτη παρατήρηση για το θέμα της συνολικής προσέγγισης. Μέσα σε αυτό το εξάμεινο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα περιεχόμενο στην έννοια της συνολικής αντιμετώπισης. Είναι κάτι που το λέμε όλοι, το τονίζουμε όλοι. Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια σημαντική χρονική στιγμή συζήτηση, όλοι περιμένουμε ακόμα την κυρία Άστο να μας πει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συνολική προσέγγιση και πώς θέλουμε να δουλέψουμε για κάτι τέτοιο. Τέταρτο, για μένα το πιο προβληματικό είναι η πολιτική θέληση, μάλλον η απουσία πολιτικής θέλησης. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει αυτή η πολιτική θέληση. Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι για τα περισσότερα κράτη-μέλη και αυτό και γενική, το γενικό κλίμα στο Συμβούλιο. Θεωρούν ότι το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με, στο πιο χαμηλό επίπεδο, θα συζητήσει λεπτομέρειες, τεχνικά ζητήματα, αλλά όχι το κεντρικό θέμα. Υπάρχει λοιπόν γενικευμένη απεσιοδοξία για τα θέματα αυτά, όταν μιλάω με τους διάφορους ε, εμπλεκόμενους στα κέντρα αποφάσεων. Για μας λοιπόν το Συμβούλιο αυτό θα πρέπει να είναι πραγματικά φιλόδοξο. Και αυτό δεν είναι μόνο η προσωπική μου άποψη, αλλά η άποψη των, των περισσότερων μελών του Κοινοβουλίου, ότι θα περνόμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και στο επίπεδο αυτό. Συμφωνούμε σε πολλά σημεία με την Κομισιόν, πρέπει να είμαστε πραγματικά φιλόδοξοι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις και το θέμα είναι πώς θα τοποθετηθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενώπιον αυτών των προσδοκιών και προ... προκλήσεων, αλλά η έκθεση του Κοινοβουλίου θα προσπαθήσει να δώσει τη δική μας άποψη και τη δική μας θέση για όλα αυτά τα αμυντικά θέματα. Επιπλέον, πρέπει να τονίσω ότι μας δίνει τα εργαλεία για να προχωρήσουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Θεσμικά. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει από τη συνήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται. Η μόνιμη διαθροντική συνεργασία, του χάρη. Για ορισμένου αυτό αφορά μόνο τη βιομηχανία. Όπως είπε και ο κύριος Μισηρόλη. Τα είπε και νομίζω πολύ εύστοχα. Έχουμε τώρα νησίδες μονάχα συνεργασίας. Η έννοια της δομικής και μόνιμης συνεργασίας θα πρέπει να αποκτήσει ένα σαφές περιεχόμενο και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Η, δική μου ιδέα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής θα πρέπει να προχωρήσουν με πιο γρήγορα βήματα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε παντού και οι 28 μαζί. Αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα θα πρέπει να έχουν τη θεσμική δυνατότητα να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μας δημιουργεί προβλήματα από αυτή την έποψη. Έκτο σημείο. Μπορούμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό της άμυνας, όχι. Αυτό αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Εμείς ως Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να προτείνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι δυνατό. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε αντίθετα είναι να βρούμε ευφυείς μεθόδους για να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους. Με την συνένωση των προσπαθειών σε ορισμένου τομεί και των ικανοτήτων. Συζητώντας με διάφορα κράτη-μέλη, λένε όλοι ότι μπορούμε να βάλουμε από κοινού τις ικανότητάς μας, αλλά το να τις διαμοιραζόμαστε και να τις χρησιμοποιούμε από κοινού, αυτό είναι δύσκολο γιατί απαιτεί μια προηγούμενη δημιουργία εμπιστοσύνης. Υπάρχουν όμως τρόποι να προχωρήσουμε προς μια πιο ευφυά άμυνα. Και υπάρχουν και τρόποι να αναδιαθρώσουμε τη ζήτηση για τα μέσα αυτά. Γιατί η αμυντική δραστηριότητα διατηρεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Εν κατακλείδη. Η έκθεση του Κοινοβουλίου είναι μια μεγάλη πρόκληση. Εφέτος, Η περισσότερη κοινοβουλευτική ανεξάρτητα από πολιτική ομάδα είναι πεπισμένη ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Άμυνας θα πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει γενική συμφωνία, αλλά αυτή είναι η πλειοψηφία. Ελπίζω ότι η Ολομέλεια του Νοεμβρίου, όταν θα ψηφιστεί αυτή η έκθεση, θα μπορέσει να δώσει ένα σαφές μήνυμα, ένα ισχυρό και στεναρό μήνυμα στο Συμβούλιο Άμυνας. Και εδώ πρέπει να είναι σαφής και ακουστή η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία και Thank you very much, Chairman. Um... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα πολλές φορές. Παραμένει το γεγονός ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τις ικανότητες και τους στόχους των ένοπλων δυνάμεων καθώς ε, και την διασφάλιση της επιβίωσης και της μελλοντική επιτυχίας των επιχειρήσεων αυτών στις χώρες μας. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση. Αν οι συνάδελφοι σε αυτή την Επιτροπή αλλά και αλλού είναι ειλικρινείς, θα αναγνωρίσουν ότι το θέμα αφορά το δεύτερο σκέλος, όχι το πρώτο. Αφορά δηλαδή την ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση. Όταν παραθέτουμε όλους τους λόγους ε, για τους οποίες δεν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέρος σε αμυντικές δράσεις, ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και το θέμα της προσέλευσης στα συμβούλια του ΝΑΤΟ, καταλάβαμε ότι λέει πολλά από μόνο του. ό,τι φορά τη βιομηχανική πλευρά, παραμένει το γεγονός ότι έχουμε πολύ επιτυχή πολλά επιτυχή προγράμματα στέφονται από επιτυχία όταν εφαρμόζονται από δύο χώρες. Είναι λιγότερο αποτελεσματικά αν συμμετέχουν πέραν των δύο χωρών. Αν έχουμε τέσσερις ή πέντε χώρες που έχουν χρήσιμες, θα λέγαμε, αμυντικές μηχανίες και εμπλέκονται στον τομέα της έρευνας. Εκεί που χρειάζεται, βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις ε, χρειάζονται κοινά προγράμματα, Typhoon, ε, Eurofighter, ε, Eurocopter, 400. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια προγράμματα. Αυτό που δεν απαιτείται εδώ είναι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει κανέναν οποιοδήποτε ρόλο να διαδραματίσει σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, αν θα μπορούσαν να συγχαρώ τους ε, συναδέλφους για το έγγραφο αυτό, το οποίο συνέταξε ο καθηγητής Κιθ ε, Χάλτρι, που είναι ειδικό στο τομέα των οικονομικών της άμυνας. Ε, ο τίτλος της ομιλίας είναι οι ελέφαντες, δηλαδή ε, ανεπιθύμητα δώρα στον τομέα της αμυντικής ε, βιομηχανίας. Στην ουσία εμείς βρισκόμαστε εδώ για ένα συγκεκριμένο λόγο και η προσπάθεια που καταβάλουμε είναι να κινηθούμε προς μία κατεύθυνση. Μενοί από εμά ε, δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό που θα μπορούσαμε να πράξουμε για το μέλλον. Πολλοί αποδίδουν σημασία στα έθνη, στις χώρες και για τον λόγο αυτό έχουμε μία εντελώς διαφορετική προοπτική ω αυτά, ως αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ των συμφερόντων για την άμυνα με τις φιλοδοξίες που έχουν για την ευρωπαϊκή ε, πολιτική ολοκλήρωση. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την αρχή της ε, παρουσίασης. Αυτό είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και εγώ προσβλέπω στην δυνατότητα συνεργασίας με τη Μαριλένα και τους κοιόδης συγητές για την έκθεση αυτή να τονίσω και δεν απαντώ εδώ στον Τζέφρι Φαν Όρντεν αλλά αν σταθώ σε αυτά που είπε εντάξει ας αφήσουμε στην άκρη όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με πολιτική ολοκλήρωση μπορείτε να φανταστείτε μια αποτελεσματική ικανότητα αμυντικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη σήμερα ότι είναι σε επίπεδο που μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ναι, λέει ο Τζέφρι, μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί αυτές είναι ικανότητες που μπορούν να επιτευχθούν μοναχά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μα θέτετε ένα ερώτημα, να απαντήσω λέει ο Τζέφρι μονομερός, ναι, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν την ικανότητα αυτή. Και ναι, από κοινού πολλά πράγματα μπορεί να κάνει η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουν από κοινού. Έχουμε και την οργανωτική δυνατότητα για, δι... για διεθνείς παρεμβάσεις που λέγεται ΝΑΤΟ, λειτουργεί πολύ καλά, χρησιμοποιεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσει την ασφάλεια της Ευρώπης και υπάρχει ένα τραπέζι στο οποίο μπορούμε να συζητούμε όλοι μαζί για την αντιμετώπιση κρίσεων και λέγεται ΝΑΤΟ. Όλα τα άλλα είναι προσώψεις και βιτρίνες. Ο κύριος ε, Βανόρντεν αυτός κάνει αυτή την άσκηση δημιουργίας βιτρινών γιατί κάναμε μια συζήτηση πρόσφατα για το ΝΑΤΟ και είχε κάνει μια πολύ σαφή πρόσκληση ο ίδιος ο κύριος Φανόρντεν στους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να κάνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ γιατί ο μόνος τρόπος να επιτευχθούν όλα αυτά είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος και αυτό το έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι αλλά ο κύριος Φανόρντεν δεν το καταλαβαίνει. Και πρέπει λοιπόν να το κατανοήσουμε αυτό. Ο μόνος τρόπος για μας να μπορέσουμε μεμονωμένα ή συνολικά να δημιουργήσουμε τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας από τις απειλές που υπάρχουν σε επίπεδο ασφαλείας περιφερειακά και παγκόσμια είναι με το να συνεργαστούμε ευρωπαϊκά να ενσωματώσουμε τις προσπάθειές μας και στον τομέα της άμυνας περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χώρο. Αυτό απαιτεί πολιτική ολοκλήρωση. Ο κύριος Φανόρντεν εκτός μικροφώνου. Όχι Τζέφρι, δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί σου. Αλλά θέλω να τονίσω ακριβώς αυτό, ότι αυτό που περιμένω από αυτή την έκθεση είναι ότι πράγματι θα δώσουμε ένα σαφές και ομό και απερίφραστο μήνυμα, όχι μόνο στις κοινέ μας γνώμες, αλλά και στις κυβερνήσεις μας ότι δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Και ότι η κρίση, η οικονομική κρίση θα πρέπει να είναι ένας περαιτέρω λόγος να προχωρήσουν σε περισσότερη ενσωμάτωση στην θέση από κοινού των εργαλείων που έχουμε και με το να μην δρουν ουσιαστικά αποτυγχάνουν να κάνουν αυτό το οποίο απαιτούν από αυτούς οι πολίτες. Θα το πούμε λοιπόν ομά και χοντρά. Πρέπει να τονίσουμε το κόστος της μη ύπαρξης της Ευρώπης, οικονομικά και μη οικονομικά. Και πάλι να τονίσω για την περίπτωση της Λιβύας, Λιβύης, συγγνώμη, όπου η κατάσταση επιδεινώνεται Κατά τη δική μου άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Η στρατιωτική παρέμβαση ορισμένων κρατών μελών με το ΝΑΤΟ δεν πέτυχε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει τώρα και τώρα δεν μπορεί να κάνει πάλι αυτό που είναι πιο σημαντικό, λιγότερο σημαντικό ή εξίσου σημαντικό να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους ε, Λίβιους για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια που χρειάζεται, όχι μόνο τη δική τους ασφάλεια, αλλά και τη δική μας ασφάλεια. Γιατί δεν μπορέσαμε λοιπόν ποτέ να έχουμε μια σωστή αποστολή άμυνας και ασφάλειας παρά τις αιτήσει των αρχών της Λιβύης για να έχουμε μια σωστή ε, διαδικασία εξασφάλισης της ασφάλειας στην ε, Λιβύη. Έχουμε μόναχα μια αποστολή για την ασφάλεια των συνόρων, αλλά εδώ εμπλέκονται πολύ περισσότερα θέματα. Είναι η πραγματική επανεκπαίδευση και μεταρρύθμιση του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας και της αστυνομίας. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Όλα αυτά γίνονται κάποια κράτη-μέλη, ιδίως αυτά που έχουν μεγαλύτερες ικανότητες, να έχουν τους δικούς τους συμβούλους κοντά στον Υπουργό Εσωτερικών της ε, Λιβύης, όπως έκαναν και την εποχή του Καντάφη, ή τουλάχιστον προσπάθησαν, ώστε να πουλήσουν το δικό τους στρατιωτικό εξοπλισμό. Και για αυτό το λόγο δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική στα θέματα αυτά, δεν υπάρχει μια κοινή προσέγγιση της Λιβύης, για να πουλήσουν κάποιοι τον εξοπλισμό τους. Είμαστε στην ίδια κατάσταση όπως την εποχή του Καντάφη που προσπαθούσε η Γαλλία να πουλήσει τα πυρηνικά της εργοστάσια των Καντάφη. Δεν μας πρέπει πουθενά αυτό. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο μη ευρωπαϊκό. Είναι κάτι το οποίο στρέφεται κατά των συμφερόντων ασφαλείας μας. Δεν μιλάει για τα οικονομικά μας συμφέροντα. Στην περίπτωση της λυφής ξέρω ότι υπάρχει πραγματική αίτηση από τις αρχές της Λιβύης για μια στρατηγικά οργανωμένη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλιστεί η μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας. Εμείς δεν το κάνουμε γιατί καποια κάποια κράτη-μέλη που τους ενδιαφέρει να επανεθνικοποιήσουν τα θέματα βιομηχανίας και άμυνας και να προωθήσουν τη δική τους βιομηχανία και τα δικά τους συμφέροντα δρούν σε βάρος των συλλογικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Με τον τρόπο αυτό λυπάμαι. Εμείς αυξάνουμε την ανασφάλεια για τους εαυτούς μας και για τους γειτονές μας. Δεν κάνουμε τα απαραίτητα. Θα σταματήσω εδώ πέρα λοιπόν. και προσβλέπω στο να συνεργαστώ περισσότερο με την Μαριλένα και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ομή γλώσσα. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θέλω να σας πω ότι ήταν ε, μεγάλη χαρά για μας το τον ακούσουμε την άποψή σας ε, και θα ήθελα να πω ότι η ανάλυση της ΕΚΕΠΑ θα πρέπει να λάβει χώρα στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προσπαθειών για να υπάρχει μια συνεπής στρατηγική προσέγγιση. Τώρα, όσον αφορά την συνένωση των προσπαθειών, το pooling and sharing, η βελτίωση στον ε, στο χώρο των επιχειρήσεων. Ε, όλα αυτές οι έννοιες απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία και εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ε, κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Ορισμένες από τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στη συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και προσφέρουν τα εργαλεία για να διευκολύνεται η ολοκλήρωση. Και επίσης ε, θεωρώ ότι ένα από τα εργαλεία που προσφέρουν προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας, οι μόνιμες δομές. Αυτές ε, είναι πολύ χρήσιμες δομές, οι οποίες καλύπτουν τα κριτήρια για την ανάπτυξη στρατιωτικών ε, δυνατοτήτων σε επιχειρήσεις. Και θέλω να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να, επιταχυνθούν, να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας, αν ναι, μπορεί να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τη σχέση ανάμεσα στο άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 5 του, της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Το 42-7 προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να προσφέρουν βοήθεια ε, σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση στο έδαφος μιας, ε, ενός άλλου ε, κράτους μέλους. Και εδώ επίθεση τι, στρατιωτική ή άμυνα. Αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 5. Και ε, το ερώτημα είναι ποιες είναι οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας ε, και κατά πόσον θέλει να γίνει κοινότητα άμυνας. Και η τρίτη μου ερώτηση είναι ε, σχετικά με τις νέες απειλές. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική έχει την δυνατότητα να μετατραπεί σε κάτι άλλο πέρα από ένα απλό χαρτί. Καταρχά να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας και για τις ολοκληρωμένες τοποθετήσεις σας και θα ήθελα να καταθέσω και το δικό μου ερώτημα αναφορικά με τα όσα έχετε ουσιαστικά εκφράσει συμφωνώντας με το έκτο θα έλεγα στοιχείο το οποίο έχετε καταθέσει ότι η άμυνα είναι καθοριστική και αποτελεί ασφάλεια για όλους μας. Σε αυτό δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει. Όμως, στον τομέα των επιχειρήσεων εκφράσετε μια υπεραισιόδοξη, θα έλεγα, τοποθέτηση και έχετε κάνει αναφορά ότι κάθε φορά που υπήρξε επιχείρηση ήταν επιτυχημένη το κατανοώ ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία, όμως η δική μου αίσθηση και εκτίμηση των πραγμάτων είναι ότι υπάρχει ένα κενό και ένα πολιτικό έλλειμμα στο θέμα των επιχειρήσεων. Ήδη συμφωνώ με την τοποθέτηση της κυρία Γκόμες που ανέδειξε το ζήτημα της θα έλεγα αποτυχία στην Λιβύη Σήμερα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Συρία όπου σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Η παρέμβαση είναι τουλάχιστον ελληματική παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Άστο και βέβαια δεν νομίζω να λύσαμε το πρόβλημα στο Μαλί, στο Αφγανιστάν ή σε άλλες χώρες. Δεν θέλω να περάσω μήνυμα απεσιόδοξο, θέλω να περάσω μήνυμα ότι υπάρχουν τεράστια, θα έλεγα, ζητήματα τα οποία πρέπει να επιτύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρώτο είναι η αύξηση βεβαίω των δαπανών που δεν φαίνεται να επιτυχάνεται ή κάποιες χώρες να μην θέλουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή πολλές φορές αλλά κάρτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ενιαία η συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Και το τρίτο, εκτιμώ ότι πέρασε ένα μήνυμα δικαίως αδίκως ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε όταν εφαρμόζουν ή αποφασίζουν να κάνουν επιχείρηση είναι αποτελεσματικοί, ενώ όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να κανουν επιχειρηση ειναι αποτελεσματική, επιχείρηση μπορεί να είναι αποτελεσματική, αλλά όχι πάντα. Ευχαριστώ. και βεβαίως μετά από τον κύκλο των ερωτήσεων το λόγο τον έχετε όλοι οι ομιλητές από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουμε χρόνο μέχρι τις μία η ώρα η παράκληση είναι να καταμεριστεί ο χρόνος 7 λεπτά για τον καθένα για να μπορέσουμε να κλείσουμε. Κόλεμα. Merci bien. Euh. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για, τις, ε, για τους προβληματισμούς που διατυπώσατε. Ευχαριστώ κυρία Κοπά. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι ένα από τα δύνατα σημεία της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας είναι το θέμα της επικοινωνίας. Έχουμε καταγράψει πολλές επιτυχίες ήδη με μια σχετική βαχύτητα, αλλά κανένας δεν τα γνωρίζει όλα αυτά. Θυμάμαι ότι πριν από την επιχειρήση στον Ταρφούρ αναπτύξαμε δράση στο υπήρξε ε, η Κομισιόν κατέβαλε την τα έξοδα όλων των Αφρικανικών στρατευμάτων. Πάρα πολύ μεγάλη στήριξη για πρώτη φορά. Μιλήσαμε για το θέμα αυτό στον τύπο. Και το θίξαμε όταν το ΝΑΤΟ έστειλε μερικά μεταφορικά αεροσκάφη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ τίθεται, υπάρχει ένα στοιχείο αδυναμίας σε επίπεδο επικοινωνία. Διαπίστωσα ότι κατά τη διάρκεια των εκλογών οι πολίτες στις διάφορες χώρες, οι πολίτες γνώρισαν <clears throat> την Ευρώπη αυτή της άμυνας. Ήταν και μία λανθασμένη αντίληψη ότι η Ευρώπη γείτο εθνικών στρατευμάτων παίρνοντα μέρο σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ένα λανθασμένο λοιπόν μήνυμα. Πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να επανορθώσουμε. Υπογραμμίσατε και άλλα στοιχεία, την πολιτική βούληση, το κοινό όραμα που μας λείπει. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μας να αναπτύξουμε μία γενική στρατηγική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για πολιτική ασφάλεια, όχι στρατηγική. Πρόκειται για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια των πολιτών, για την ασφάλεια όσων μας περιβάλλουν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε αυτό να γίνει ένα έγγραφο ελκυστικό, μια ελκυστική αφήγηση. Στο παρελθόν έγιναν πόνοι και πόλεμοι, αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε με μία ήπειρο. Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο μίας ήπειρου που θέλει να προασπίσει όχι μόνο τα δικά της συμφέροντα και τις αξίες αλλά να αποτελέσει και ένα σημαντικό παράγοντα με προστιθέμενη αξία σε επίπεδο παγκόσμιο και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιδιώξουμε μια καλύτερη επικοινωνία. Κύριε Βανέντεν, θυμάμαι ότι πριν από ένα χρόνο καθόμουν εδώ και μου κάνατε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Σας έδωσα μία απάντηση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν σας έπεισα. Το σημειώνω. Κυρία Γουμάσα, πιστεύω ότι αυτό που βλέπει η Ευρώπη είναι ότι δεν έχουμε όλοι μια κοινή άποψη για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τον, την εθνική αντίληψη, η οποία μας οδηγεί στις καταστάσεις που περιγράψατε. Αυτό που αποτελεί απάντηση και σε αυτό που είπε ο κύριος ε, Πανέτα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Στρατηγική είναι ένα έγγραφο όπως όλα τα έγγραφα. Τα έγγραφα μας περισσεύουν. Αυτό που μας λείπει είναι μια πραγματική στρατηγική. Η στρατηγική είναι μια αντίληψη, μια νοοτροπία, όχι ένα κομμάτι καρτί. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα κατανοήσουν αυτή τη στρατηγική. Αυτό που λέω είναι ότι ο τρόπος έχει την ίδια βαρύτητα με το αποτέλεσμα. Οι χώρες θα πρέπει να έχουν άμεση συμμετοχή. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ κρατών και κυβερνήσεων. Πολύ συχνά αφορούν καταστάσεις όπως αυτή στο Μαλί. Στο Ε, ποτέ δεν συνειδητοποίησαν οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων τη στρατηγική που αναπτύχθηκε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σαχάρα, στο κέρας της Αφρικής. Καταλαβαίνετε ότι <clears throat> δεν συνειδητοποιούν οι επικεφαλείς κρατών ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι το ανακαλύπτουν, δεν καταλαβαίνουν την υποχρέωσή τους να κάνουν κάτι στα πλαίσια μιας κοινή στρατηγικής. Δεν θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό δεν είναι μια απάντηση στα περισσότερα ερωτήματα και πρωτίστως το ερώτημα πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ανεπάρκειές μας. Ε, ή θα συμπορευτούμε ή θα πορεύεται ο καθένας μόνος του. Με τους κινδύνους βεβαίως που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το στοιχείο αυτό για το άρθρο 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 5 των Ηνωμένων Εθνών, έχω τη χαρά να δίνω διαλέξεις στα πανεπιστήμια και όταν δίνω ενώπιον ε, φοιτητών της νομικής ε, σχολής τονίζω ότι υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο άρθρων. Δεν είναι ταυτόσιμα αυτά τα άρθρα. Όταν ε, μιλάω στην ε, Σχολή Πολιτικών Επιστημών, τότε στην αυτή περίπτωση δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και από την πολιτική και στρατιωτική μου εμπειρία θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά μεταξύ των δύο άρθρων. Κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια για τα ερωτήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε η κυρία Κοπά. Πράγματι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε επίπεδο επικοινωνίας γιατί φαίνεται ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τα πράγματα καλύτερα πολλές φορές και εδώ σας υποστηρίζω. Πολλοί καταλαβαίνουν πόσο δύσκολες είναι οι εποχές που αντιμετωπίζουμε, πόσο χαλε, χαλεπή η καιρή σε επίπεδο ασφάλειας, σε παγκόσμιο επίπεδο και στρατηγικά και οικονομικά. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία για τα θέματα αυτά και καλύτερη αντίληψη και συνειδητοποίηση. Το ΝΑΤΟ κάνει μια άσκηση επικοινωνίας που λέγεται Defense Matters η οποία θα περατωθεί το φθινόπωρο και έχει ακριβώς σαν στόχο να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Για τον κύριο Φανόρντε. Νομίζω ότι έχετε αντιμετωπίσει με λανθασμένο τρόπο τη συζήτηση. Την διατυπώνετε με τρόπο που λέτε εδώ βρισκόμαστε, λέτε, για να βρούμε ένα άλλο τρόπο να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όχι, η δική μου αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Ο στόχος συζήτησης είναι να μείνει η Ευρώπη ευμαρής, ειρηνική και ελεύθερη. Είτε το πετύχει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ τελικά δεν έχει καμιά σημασία. Συμφωνώ μαζί σας ότι προς το παρόν το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή και μάλλον στο ορατό μέλλον θα είναι αυτός ο οποίος θα φέρει αυτές τις υπηρεσίες ασφάλειας. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται πάρα πολύ από την θέληση των Αμερικανών να το εξασφαλίσει αυτό και όχι από τους Ευρωπαίους όπως είναι τώρα τα πράγματα. Το να εξαρτιόμαστε μόνο από τους Αμερικανούς μπορεί να είναι πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι αδύρυτο να είναι πρόβλημα, αλλά ο πραγματικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την ευμάρια ασφάλεια και ελευθερία της Ευρώπης. Το να μην χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους θα είναι λαθασμένο. Έχουμε δύο παρόχους ε, υπηρεσιών ασφάλειας. Το ΝΑΤΟ είναι ο τωρινός πάροχος, η Ευρώπη είναι ένα δευτερεύον εργαλείο, αλλά με πολλές προοπτικές θα ήταν λαθασμένο να μην το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Δεν θέλω λοιπόν να πω ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας μπαμπούλας που θέλει να προωθήσει περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά δεν μπορούμε να ξεφτόμαστε για πάντα από τις ΗΠΑ. Για αυτά που είπε η κυρία Παναγιώτοβα. θέσατε αυτά τα ερωτήματα για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να γίνει μια δύναμη σε επίπεδο ασφάλειας. Όχι, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε κάποιο επίπεδο ασφάλειας. Μια κοινότητα ασφαλείας, όχι μόνο με την έννοια του άρθρου 5, αλλά με την έννοια ότι είμαστε στην Ήπειρο αυτή όλοι μαζί και έχουμε κοινά συμφέροντα και μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό που έχει αναφερθεί από ορισμένους ανελτές όσον αρκεί των μικρών διαφορών. Υπάρχουν διαφορές, αλλά οι διαφορές αυτές είναι πολύ μικρές σε σχέση με το γενικό πλαίσιο. Αν ξεπεράσουμε λοιπόν αυτές τις διαφορές, υπάρχουν κοινοί στατιστική στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι, Ευρωπα... οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Και γι' αυτό εγώ πράγματι υποστηριζώ να τα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δεύτερο ερώτημα σας αναφερθήκατε στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τέτοιο ερώτημα όπως εμάς για το θέμα αυτό. Αλλά μπορούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από μια χάρτινη τίγρη. Αυτό είναι πάντα το ερώτημα. Ε. Τα κράτη-μέλη αν έχουν μια πολιτική η οποία είναι αποσπασματική για τα θέματα ασφαλείας δεν θα επιτύχουν το στόχο αυτό. Υπάρχουν κάποιες χρήσιμες ιδέες, η πιο σημαντική η αξία του εγγράφου μας. Το ξαναλέω αυτό συνέχεια σαν μία μάντα. Είναι ότι υπάρχουν κάποιες αναγκαιότητες πρέπει να τις αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελική μου παρατήρηση για το άρθρο 5 είναι ένα παράξενο ζώο το άρθρο 5. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι το άρθρο 5 ακόμα και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου δεν σήμαινε πολλά πράγματα. Η εγγύηση ασφάλειας του ΝΑΤΟ δεν προερχόταν από το άρθρο 5, αλλά από το γεγονός ότι κυρίως το γερμανικό έδαφος αλλά και αλλού ήταν παρόντα τα στατέματα όλων των κρατών του ΝΑΤΟ. Οι Καναδοί, οι Αμερικανοί, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, οι Έγγλοι Επομένως μια επίθεση στο γερμανικό έδαφος θα ήταν μια επίθεση εναντίον όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η πραγματική εγγύηση. Το άρθρο 5 είναι απλώς μια διάταξη στην συνθήκη του ΝΑΤΟ. Και είναι το αντίστοιχο με το άρθρο 42 στο Ευρωπα... στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Το θέμα είναι από πού προέρχεται η πραγματική αλληλεγγύη. Έρχεται από παρουσία στρατευμάτων επιτοπίως ή από μια συνείδηση του ότι πρέπει να παραμείνουμε μαζί για μένα δεν φτάνει πια η παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος. Η αλληλεγγύη προέρχεται από τη συνειδητοποίηση ότι υπάρχει μια κοινή απειλή και ότι είναι πια τα κοινά μας συμφέροντα στον κόσμο και ξεπερνούν πια τα στρατιωτικά θέματα. Είμαστε μια περιοχή που βασίζεται στο εμπόριο, έχουμε έλλειψη εργατικών δυνάμεων και δεν έχουμε βασικούς πόρους. Μας συνδέει το κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της παγκόσμιας οικονομίας. Αν λοιπόν αυτό δεν οδηγήσει σε αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαίων, δεν θα μας πάει πουθενά. Δεν θα έχουμε από πουθενά ασφάλεια είτε από το ΝΑΤΟ είτε από κάπου αλλού. Um, Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διχογνωμία που υπάρχει μεταξύ των βουλευτών και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η προσπάθεια που καταβάλαμε είναι να ζητήσουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων. Αυτό δεν ήταν ένα πολιτικό επιχείρημα. Το επιχείρημα βασίζεται στα δικά μας συμφέροντα, γιατί αν κοιτάξουμε το πώ έχουν τα πράγματα σήμερα, η περικοπή των αμυντικών δαπανών στο εθνικό επίπεδο, η κάθε χώρα ξεχωριστά με βάση την ισχύουσα δημοσιονομική λογική δυνητικά οδηγεί στη δημιουργία σμικριμένων στρατών, στρατών ε, bonsai. Ε, και βεβαίως οδηγεί και την ενδυνάμωση άλλων ανταγωνιστών. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε ήδη αλλού και αν δείτε τα στοιχεία που έχουμε από το Διεθνές Ινστιτούτο Ασφάλιση Στρατηγικών Μελετών στο Λονδίνο, συνειδητοποιούμε ότι το μοναδικό μέρος του κόσμου όπου οι δαπάνε, οι αμυντικές δαπάνες συστηματικά μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι η Ευρώπη. Βλέπετε όμως ότι αλλού είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αύξηση στον τομέα των δαπανών. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες αγορές. Και το βασικό επιχείρημα που προσπαθούμε να προβάλλουμε είναι ότι είναι πιο αποτελεσματική η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυνητικά, γιατί δεν έχουμε δει μέχρι στιγμή και πολλή συνεργασία. Ή διμερός, ή σε εθνικό επίπεδο, ή τριμερός και αυτό για δύο βασικούς λόγους. Καταρχάς, λόγω της ικανότητας που δυνητικά έχει η Ευρώπη να ε, κινητοποιεί, ε, να χρησιμοποιεί μπορούσε ε, και αυτό το διαπιστώσαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και επίσης και θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό λόγω της συλλογικής ρυθμιστικής εξουσίας που έχει η Ευρώπη. Αυτό αφορά τις προλογικές πολιτικές, ε, γενικές δαπάνες σε, διεθνές, ε, σε εθνικό επίπεδο αλλά αυτό αφορά και τους κανόνες των προμηθειών, των κοινών προγραμμάτων, έρευνας, ανάπτυξης, ε, τεχνολογίας κτλ. Αυτό είναι κάτι που δεν διαθέτει καμία άλλη οργάνωση στον κόσμο, το κάνει το ΝΑΤΟ. Επίσης, θα σας έλεγα ότι είναι επικίνδυνο το να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα με παροπίδες. Εάν οι, <clears throat> οι Ευρωπαίοι καταφέρουν να δράσουν σε αυτό το τομέα, θα προκύψουν ωφέλη και για τον ΝΑΤΟ. Και αν καταφέρουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί, πιο καινοτόμοι, αυτό θα αποβεί υπέρ όλων. Ατλαντικής Συμμαχίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ξεκίνησε η δράση στο Λίβανο το 2006 ήταν μια επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών με επικεφαλή στην Ευρώπη. Αλλά όλοι συμφωνήσαμε ότι πολιτικά ήταν περισσότερο σκόπιμο η δράση να περάσει από τα κανάλια των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν θα είναι στην διάθεση της διεθνούς ασφάλειας. Ακόμα και αν η βασική λογική για να ε, δραστηριοποιηθούμε από κοινού είναι βασικά ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Ομπάμα δεν θα έχει αντιρρήσεις γιατί είναι εύκολο να δουν ε, τα αποτελέσματα. Είναι θέμα καθαρά πρακτικό, ιδεολογικό. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό της πολιτικής, θα επιμείνω. Δεν θα πρέπει στενόμυαλα να κοιτάμε μόνο το τομέα της άμυνας. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις ε, επιχειρήσεις. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία που συμβάλλουν εκεί. Όσο περισσότερα είναι τα στοιχεία, τόσο πιο ε, επιτυχής η έκβαση αυτών των επιχειρήσεων. Οι στρατιωτικές δυνάμεις από μόνες τους δεν είναι ο μοναδικός, η ε, ε, στρατιωτική ισχύ δεν είναι ο μοναδικός τρόπος επίλυσης των θεμάτων. Ο πολιτικός συντονισμός θα πρέπει να ξεπερνάει τα στενά όρια της άμυνας. Τα άλλα τα επιχειρήματα είναι απλώς παραπλανητικά. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε Ευχαριστούμε τους υπουργούς ε, και όλους τους παίκτες που έπαιξαν ρολό. Μία από τις απώλειες της συνθήκης Λισαβόνας είναι ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών είναι όλο και λιγότερο σημαντικοί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θεωρεί τους ε, Υπουργούς Εξωτερικών σαν μέρος της διαδικασίας. Αυτό είναι κάτι αρνητικό. Στο παρελθόν θα θυμάστε ότι πάντοτε γινόντουσαν συζητήσεις σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και στα συμπεράσματα συνεπάγεται ε, και ε, στα συμπεράσματα συνεπολογιζόταν και η δική τους άποψη και υπήρχε ένα στοιχείο εξωτερικής πολιτικής. Ε, η τελευταία συζήτηση για τέτοια στρατηγικά ε, θέματα έγινε το 2008 κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας. Έγινε μια προσπάθεια για επανάληψη αυτών των συζητήσεων το 2010 και μετά την πρωτοκαθεδρία την είχαν τα στρατηγικά θέματα. Συνεπώς ε, επαναλαμβάνουμε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να έχουν άποψη. Γιατί όταν τίθεται θέμα ε, καταμερισμού των πόρων θα πρέπει και εκείνοι να κατανοήσουν τις στρατηγικές προτεραιότητε, όπως και άλλοι θα πρέπει να κατανοήσουν τις ε, προτεραιότητε του προπολογισμού. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα στο μέλλον. ενδεχομένω. θα θυμάστε ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε το Συμβούλιο Μαμούθ, όπου συμμετείχαν οι Υπουργοί Άμυνα, Αναπτυξιακή Βοήθεια και Εξωτερικών. Ενδεχομένω μπορεί να έχουμε αντίρρηση ε, στην επωνυμία. Το μαμούθ είναι ζώο μεγάλο και ζώο που πλέον έχει εξαφανιστεί. Θα μπορούσαμε όμως να βρούμε μια ε, ε, δημιουργική λύση σε αυτό το επίπεδο. Αν θέλουμε να του δώσουμε ένα όνομα, σώνει και καλά, γιατί όχι καμιλοπάρδελη. Καμιλοπάρδελη είναι ένα δόζο ευκίνητο με τα πόδια στη γη, ζει στην Αφρική, ας το έχουμε και αυτό στο νου μας, είναι ένα ζώο που βλέπει ψηλά, βλέπει μακριά γιατί έχει ψηλό λαιμό και δυνητικά μπορεί να τρέξει. Γιατί η καμιλοπάρταρης μπορεί να αναπτύξει πραγματικά εγκυπωσιακή ταχύτητα. Κύριος Μαρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να φέρω μία σειρά θεμάτων. Μερικά θέματα. Η ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας. Ναι. Όπως προσπάθησα να πω στην παρουσίασή μου, τα θέματα του αμυντικού τομέα δεν είναι μόνο η ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά είναι και η τεχνολογική καινοτομία, οι τεχνολογίες διτής χρήσης, εξαγωγές. Είναι επομένως η βιομηχανική ικανότητα, η διατήρηση της βιομηχανικής ικανότητας στην Ευρώπη είναι τελικά η οικονομία. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι οι μόνιμες δομές συνεργασίας, όπως ανέφερε η κυρία Παναγιώτοβα. Η εξέταση των δυνατοτήτων συνεργασίας είναι πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάτι μέλη που θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα, να μπορέσουν να δράσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως, είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά ανοιχτή και διάφανη. και ενσωματωμένη στο θεσμικό πλαίσιο για να μπορούν και άλλα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή τη μόνιμη συνεργασία ή να έχουν μια ευέλικτη σχέση με αυτή. Εξισορροπεί λοιπόν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευκαμψία με την ανάγκη να μην υπάρξει κάποια διαταραχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Για την Λιβύη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στη συζήτηση, να είμαστε σαφείς. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έκανε τις περισσότερες επιχειρήσεις κρούσεως τις πρώτες μέρες. Ήταν η υψηλότερη τεχνολογία και οι πιο ρισκαρισμένες επικίνδυνες επιχειρήσεις στους επόμενους 7 μήνες της αεροπορικής επιχείρησης δεν έκανε παραπάνω από το 1 τρίτο κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από το 1 τρίτο των πτήσεων πάνω από τη Λιβύη. Επομένω, καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν μπορεί μόνη της να κάνει μια επιχείρηση όπως αυτή της Λιβύης. Ακόμα και δύο χώρε θα το βρουν δύσκολο, αν όχι αδύνατο να διαχειριστούν μια τέτοια επιχείρηση. Τέταρτη παρατήρηση, η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εμείς εμπλεκόμαστε και ο οργανισμός στον οποίο συμμετέχω για τη στρατηγική αυτή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο στόχος ήταν να δώσουμε ένα έναυσμα στη συζήτηση και σε τελική ανάλυση όλα αυτή η εκτιμένη δράση, αν υπάρχει πολιτική θέληση, αλλά κυρίως η πολιτική συνειδητοποίηση όλων αυτών των προβλημάτων, της ανάγκης να έχουμε μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και δράση. Και εδώ το γεγονό ότι, όπω είπα προηγουμένω, δεν υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή χώρα η οποία μπορεί να φέρει σε πέρα μια επιχείρηση όπω αυτή τη Λιβύης Και το γεγονό ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αεροδιαστημικού χαρακτήρα και άμυνα εξαρτάται από κάποιε ευρωπαϊκέ δράσει. Όλα αυτά μα δείχνουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η πολιτική συνειδητοποίηση της ανάγκης να υπάρξει μια ευρωπαϊκή δράση για τα θέματα άμυνας. Τέλος, θέλω να πω ότι μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, που είναι απαραίτητη για το λεγόμενο pooling and sharing, το να θέτουμε από κοινού τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φτάνει πια στα όρια του αυτό το σύστημα, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα, μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων, χωρίς να υπάρχει και μία εκ των άνω προς τα κάτω κίνηση από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με την ενοποίηση της, των αμυντικών προμηθειών και την ορθολογικοποίηση σε ό,τι αφορά την πολιτική βιομηχανίας για τον αμυντικό τομέα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φιλοξενούμενους μας και η ώρα 3 συνεχίζουμε την κατάσταση του ευχαριστά.